Good. Meine Damen und Herren. Πολύ καλά κύριε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα έλεγα να ξεκινήσουμε. Ακόμα και αν ο συμπρόεδρος, η κυρία Βαλενσιάνο δηλαδή, δεν παρίσταται. Αλλά θα προσέλθει εντός ολίγου. Αλλά επειδή έχουμε περιορισμένο χρόνο, να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις εργασίες μας. χαίρομαι που σήμερα έχουμε αυτή την ακρόαση από κοινού με την Αλκοινοβουλευτική Επιτροπή για τα θέματα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και το, τους όρους υπό τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίζονται στις περιφερειακές συμφωνίες εμπορίου και ιδιαίτερα σε σχέση με τις αφρικανικές χώρες. Θα ήθελα να σας καλοχαιρετήσω όλους σας θερμά τους συναδέλφους φυσικά πρώτα, αλλά και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και όσους μας παρακολουθούν από την επιστήμη και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Και θα χαιρόμουν για το ότι έχουμε τέσσερις επαΐοντες παρόντες που θα μας επεξηγήσουν όλα τα σχετικά θέματα. Τον καθηγητή Γιάνν Βόρτος πρώτα. Καλώς ήρθατε που νομίζω μια ευρύτατη ανάλυση έχει εκπονήσει και στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος για την έρευνα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε βάθος έχει εργαστεί και έντονα και τον κύριο Λότζ επίσης θέλω να καλωσορίσω σε σχέση με την παρουσία του καλώς ήρθατε τον κύριο Τζάγκες Κοντιούλ, που είναι ο, πρόεδρος, ο πρέσβης του Μαυρικίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εσείς καλώς ήρθατε πρέσβη και τον κύριο Ζακ Μπερτελό έναν επιστήμονα για τα αγροτικά θέματα της μη κυβερνητική οργάνωσης από την Γαλλία Αλληλεγγύη Solidarité ένα ολόκληρο φάσμα, ευρύ φάσμα πραγματογνωμόνων που στα πιεστικά ερωτήματά μας ε, θα μπορέσει να δώσει απαντήσεις. Το πλαίσιο πρώτα να παρουσιάσουμε εισαγωγικά. Καταρχήν πρώτα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχουμε μια ολόκληρη σειρά τέτοιων συμφωνιών που θα εξεταστούν και θα συζητηθούν από κοινού με τις διαπραγματεύσεις που εδώ και πολλά χρόνια διεξάγονται με τις χώρες της Αφρικής και που εμείς ε, ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να αξιολογήσουμε και στο τέλος να επικυρώσουμε φυσικά. Οι όροι και προϋποθέσεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου που εμπεριέχονται σε αυτό το πλαίσιο είναι κάτι που έχουμε αρχικά συζητήσει μεν, αλλά δεν έχουμε τελεσίδικα ολοκληρώσει και αξιολογήσει. Τίθεται το θέμα ποιες είναι οι προϋποθέσεις και οι όροι για την Συμφωνία Κοτονού για παράδειγμα. Πώς τέτοιοι όροι και προϋποθέσεις σε τέτοιες συμφωνίες πρέπει να αξιολογούνται. Πόσο ισχυρή είναι η εξέλιξη των πραγμάτων και η ανάπτυξη αυτών των θεμάτων. Και το θέμα των δικαιωμάτων του ανθρώπου φυσικά στη δική μας ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή έχει τεράστια σημασία ως ένα θεμελιώδες στοιχείο σύγχρονων εμπορικών συνθήκων και συμφωνιών. Το είδαμε και στο πλαίσιο της GSP. Ο Ντέβιν Μάρτιν έχει εργαστεί σε βάθος για αυτά τα θέματα. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό κατοχυρώνονται και στο πλαίσιο των Delegated Acts ως ευθύνη του Κοινοβουλίου εκφράζεται με σαφήνεια. Και έχουμε και καταστάσεις σε δυτικοαφρικανικά κράτη που αν δούμε τι συμβαίνει εκεί, τίθεται το ερώτημα κατά πόσον με τέτοιες ρήτρες εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι να βελτιωθεί η κατάσταση εκεί. Ακριβώς αν δει κανείς για παράδειγμα το 80% της παραγωγής κακάου προέρχεται από τη Δυτική Αφρική για την παραγωγή σοκολάτα στην Ευρώπη, πρέπει να δούμε τι γίνεται και τι συμβαίνει εκεί με αυτή την σοδιά, σοδιά κόκκων κακάου που καλύπτεται με παιδική εργασία εκεί και πραγματικά όροι και προϋποθέσεις πρέπει να εξεταστούν για όλα αυτά τα θέματα και να καταστεί σαφές σε ποιο βαθμό εμείς μέσω τέτοιων ε, συμφωνιών μπορούμε να συνεισφέρουμε στη βελτίωση της κατάστασης στις χώρες αυτές. Αυτό αποτελεί αντικείμενο λοιπόν της συζήτησης σήμερα και χαίρομαι ιδιαίτερα που ο συμπρόεδρος, η κυρία Βαλενσιάνο δηλαδή, τώρα είναι ανάμεσά μας πλέον και της δίνω αμέσως τον λόγο για την εισαγωγή της, για τις παρατηρήσεις της. Παρακαλώ κυρία Βαλενσιάνου. Buenos días. Perdón por el... Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα, αλλά ήμουν σε μια σε μιας υποεπιτροπής και γι' αυτό καθυστέρησα. Σας ευχαριστώ καταρχάς και κυρίως τον πρόεδρο Λάγκε, τον ευχαριστώ για την πρόσκλησή του. Νομίζω ότι είναι σημαντικό και θεμελιώδες το γεγονός ότι εγκύπτουμε σε κάποια θέματα με συντονισμένο τρόπο. Και η συνεργασία μεταξύ δύο σημαντικών ε, επιτροπών, της δικής Επιτροπής ΣΥΝΤΑ και της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενισχύει τις θέσεις μας και αυτό αντικατοπτρίζεται και στην κοινή γνώμη, φτάνει ως τα κράτη-μέλη και στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν. Νομίζω ότι το να προχωρήσουμε χέρι-χέρι θα μας καταστήσει πιο αποτελεσματικούς. Η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένα σαν, σκουλίκι, κάτι που, που ενοχλεί, ενοχλεί την πολιτική ατζέντα, ενοχλεί συνειδήσεις. Είναι ένας διαολάκος αλλά αυτό, αυτή η δέσμευση αναλάβαμε απέναντι στους Ευρωπαίους. Ε, να υπερασπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα πέρα από τα σύνορά μας. Υπάρχει και μια νομική εντολή που έχει δώσει και που αναφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας. Πρέπει να το κάνουμε και οφείλουμε να το κάνουμε με ξυπνάδα, χωρίς κοινικότητα. Χωρίς κινησμό, τι σημαίνει. Ότι πρέπει μερικές φορές να παρενοχλούμε συνειδήσεις, να ενοχλούμε άλλους. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να προβληματιστούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κατάστασή τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν κάποιος υπογράψει μια συμφωνία οικονομική εμπορική με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φανταστείτε μια ανώτερη, μια ισχυρότερη δύναμη που υπογράφει ας πούμε μια συμφωνία οικονομική ή εμπορική μαζί μας. Έτσι. Και έβλεπε ότι εμείς διαλύουμε το σύμπαν, ας πούμε, τη μετανάστευση. Φτάνουν, ας πούμε, μετανάστες στην ε, Μεσόγειο, ε, πρόσφυγες κτλ. Και, και δημιουργείται χάος. Ε, αν κάποιος εξωτερικός μας έλεγε Α βάλουμε μία ρήτρα σε αυτή τη συμφωνία που θέλετε να υπογράψετε με την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση ε, την οποία ρήτρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαχειριστεί με διαφορετικό τρόπο του μετανάστε που φτάνουν στι ακτέ μα. Έτσι. Για κάτι τέτοιο μιλάμε. Μιλάμε για να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο των εμπορικών σχέσεων ω εργαλείο που θα διευκολύνει την προώθηση και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το κάνουμε. Ή δεν το κάνουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα το πρωί, ούτω ώστε οι εμπειρογνώμονε να μα εξηγήσουν εάν οι εμπορικέ συμφωνίε εξυπηρετούν αυτό το στόχο, το, την προώθηση δηλαδή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ε, Αφρικανική Ήπειρο. Και σα ευχαριστώ πάρα πολύ που μα προσκαλ, ε, προσκαλέσατε για να συμμετάσχουμε κι εμεί σε αυτή την ακρόαση. Σα ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα καταρχήν θα λάβει τον λόγο πρώτο πραγματογνώμων, ο καθηγητή, κ. Γιάνν Βάουτερ. Για 7 λεπτά έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Ε, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Κυρίες και κύριοι, μεγάλη τιμή να παρίσταμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι ο Γιάνν Βάτρος, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Λουβένης και είμαι και συντονιστής ε, ενός μεγάλου προγράμματος πλαισίου ευρωπαϊκής κλίμακας που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εξωτερικές και εσωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά από αυτά που θα σας παρουσιάσω σήμερα βασίζονται στις σημερινές έρευνες στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου. Και θα σας στείλω τις διαφάνειές μου, του PowerPoint και κάποιες από τις πρόσφατες ε, εκθέσεις μας μετά από τη συνοδοφή. Εδώ θα κάνω μια εισαγωγή και να σας παρουσιάσω το πλαίσιο των προϋποθέσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των διεθνών και περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών. Αντιλαμβανόμενοι τώρα ότι βρισκόμαστε ε, στην περίοδο μετά τη Λισαβόνα για πέντε χρόνια όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μια από τις θεμελιώδεις αξίες και θεμελιώδης στόχος της εξωτερικής πολιτικής όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης σαφές ε, όχι μόνο υπό την έννοια ότι η δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ολόκληρο τον κόσμο πρέπει να καθοδηγείται από την οικουμενικότητα και την ορθότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά επίση, διότι ακόμη πιο σημαντικό όλοι οι τομεί τη εξωτερική πολιτική πρέπει να βασίζονται σε αυτά συμπεριλαμβανομένη τη κοινή εμπορική πολιτική και των εξωτερικών συμφωνιών που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαντικό είναι επίσης ε, να αναφερθούμε στην ε, ε, χρήση της συνθήκης της Λισαβόνας μέσω του πλαισίου και του σχεδίου δράσης του 2012 για το εμπόριο, όπου προβλέπεται ότι η εμπορική πολιτική πρέπει να λειτουργεί με τρόπο τέτοιο που να υποστηρίζει τα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και όπως γνωρίζετε, ετοιμαζόμαστε να εγκρίνουμε στο Συμβούλιο ένα νέο σχέδιο δράσης του 2015 το οποίο πράγματι περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις για το εμπόριο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και πιο συγκεκριμένα ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναφέρονται στην ανάγκη βελτίωση της συνοχής όσον αφορά την εφαρμογή των ρητρών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συστηματικά συμπεριλαμβάνονται σε κάθε νέα διεθνή συμφωνία εμπορική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να διασφαλίσει τη συνοχή πολιτικής μεταξύ των διαφόρων τομέων εξωτερική και εσωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που αποτελεί συχνά μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι άλλο που είναι αρκετά σημαντικό όσον αφορά τι διεθνεί συμβάσει που συνάπτει και διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πολυμορφία των συμφωνιών. Κάποιε είναι καθαρά εμπορικέ, η FTA, Κάποιε άλλε είναι συμφωνίε εμπορική και οικονομική συνεργασία, κάποιε άλλε είναι συμφωνίε σύνδεση και κάποιε άλλε είναι αυτό που ονομάζουμε ενισχυμένε ε, συμφωνίε σύνδεση με συγκεκριμένε χώρε όπω ε, τη νότια και ανατολική γειτονία, ε, τι χώρε ACP, τι υποψήφιε χώρε και ούτω καθεξή. Γιατί είναι σημαντικό και αυτή η πολυμορφία, διότι η νομική βάση είναι διαφορετική σε ορισμένου τομεί. Έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κάποιου άλλου τομεί που αφορούν την αναπτυξιακή συνεργασία έχουμε κοινή ε, αρμοδιότητα. Πράγμα περιπλέκτα πράγματα. Υπάρχει λοιπόν πολυμορφία όσον αφορά τι συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν αναφερόμαστε στι αφρικανικές χώρε πρέπει να γνωρίζετε ότι ορισμένε τέτοιες χώρες υπόκεινται σε διαφορετικά είδη διεθνών συμφωνιών. Τι συμβαίνει όμως σήμερα. Όλες αυτές οι συμφωνίες σήμερα περιλαμβάνουν τις ε, επωνομαζόμενες ρήτρε ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν το δούμε ιστορικά, για να βρούμε πότε δημιουργήθηκαν αυτές οι ρήτρε ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, αυτές έχουν ενισχυθεί και εμφανίζονται όλο και πιο συχνά με το πέρασμα του χρόνου. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε εδώ ότι στις σημερινέ διεθνεί συμφωνίες τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι. Βάσει τη λογική ότι υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ω εργαλείο και εφόσον χρειαστεί και ως νομική βάση για την αναστολή και εφαρμογή αντιμέτρων στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών. Κάτι πολύ ενδιαφέρον, οι ρήτρε ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι επίση ε, κάτι που λαμβάνει διάφορε μορφέ. Δεν υπάρχει κάποια τυποποιημένη ρήτρα. Ε, υπάρχουν ε, διάφορα είδη, εκφράζονται με διαφορετικού τρόπου, αλλά αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι ανάλογα με το προφίλ τη χώρα και τη περιφέρεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει μια διαφοροποίηση στι ρήτρε ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίση, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι αυτέ οι ρήτρε σήμερα υποστηρίζονται από ρήτρες μη εκτέλεσης. Πρόκειται για διατάξεις εντός των συμφωνιών που προέκυψαν κάπως αργότερα χρονικά όπου υπάρχει ένας μηχανισμός παρακολούθησης, follow-up ε, για τις διαβουλεύσεις και για ενδεχόμενα κατεπήγοντα μέτρα σε περίπτωση ε, ε, ουσιαστικής παραβίασης ε, Τη συμφωνία, ε, που περιλαμβάνει φυσικά τι ρήτρε ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φυσικά το πρόβλημα με αυτές τις ρήτρε ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι απλά η πολυμορφία του και οι διαφορετικέ νομικές βάσει, αλλά και η παρακολούθηση, το follow-up δηλαδή και η πρακτική εφαρμογή, η παρακολούθηση και η επιβολή αυτών των ρητρών. Να σας δώσω, να σα παρουσιάσω δύο σημαντικά ζητήματα που έχουμε εντοπίσει στις εκθέσεις πλαίσια μας ε, ως προβληματικά όσον αφορά την αιρεσιμότητα για θέματα ανθρωπίνων δικαιωματών στις διεθνείς συμφωνίες. Πρώτα απ' όλα, έχουμε διάφορες τομεακές εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που προβλέπουν την απελευθέρωση του εμπορίου ή τη συνεργασία για ορισμένα συγκεκριμένα προϊόντα ή τομείς υπηρεσιών. Εκεί ανακαλύπτουμε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένε ρήτρε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει ένα νομικό επιχείρημα για το κατά πόσο αυτές οι τομεακές συμφωνίες πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις άλλες συμφωνίες και ετήθηκε και άλλο ένα ζήτημα το οποίο θεωρώ πολύ ενδιαφέρον αλλά περίπλοκο το ζήτημα της προσωρινής εφαρμογής των διεθνών συμφωνιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζετε πόσο πολύπλοκες είναι οι επανομαζόμενες μικτές συμφωνίες όπου υπάρχει μεικτή αρμοδιότητα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών αυτό σημαίνει ότι συχνά για ένα ή δύο έτη, τουλάχιστον αρχικά, περνάμε από το μέσο της προσωρινής εφαρμογής και αυτή η προσωρινή εφαρμογή ενίοτε λαμβάνει χώρα χωρίς να αναφέρεται στην ευρύτερη συμφωνία. Δηλαδή μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου δεν εφαρμόζεται δεν εφαρμοστεί οι προποθέσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τουλάχιστον κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογή τη συμφωνία. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπω οι πολλέ διαφορετικέ διατυπώσει των ρητρών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το γεγονό ότι σήμερα οι διεθνεί σύμφωνίε, ε, τι οποίε διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβάνουν και κεφάλαια βιώσιμη ανάπτυξη, όπου συχνά γίνεται αναφορά σε θεμελιώδη ε, κοινωνικά δικαιώματα εδώ φτάνω προς το τέλος βέβαια γιατί βλέπω ότι ολοκληρώνω το χρόνο μου. Η πραγματική ε, παρακολούθηση και το follow-up και η επιβολή των ρητρών ανθρώπινων δικαιωμάτων ε, δημιουργεί κάποια προβλήματα. Κάποιες πρώτες μελέτες παλιότερα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέδειξαν ε, έλλειψη παρακολούθησης, έλλειψη πολιτικής συνοχής. Οπότε πρέπει να επανεξετάσουμε το όλο ζήτημα γιατί τίθεται ζήτημα αποτελεσματικότητας εδώ. Τίθεται ζήτημα νομιμότητας, αξιοπιστίας και από αυτή την έννοια καλό θα ήταν να, επισημάνουμε ότι το σχέδιο δράσης του 2015 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία αναφέρεται ξανά στις συμφωνίες ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις σημερινές, για τις σημερινές και τις μελλοντικές συμφωνίες που θα συνέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ καθηγητά Βάτερς για, τα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Δίνω το λόγο στην κυρία Τζόνια Λότζ. Ähm, σας ευχαριστώ θερμά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ ενώπιόν σας και μπορώ να παρουσιάσω και να πω ότι εγώ υπό την ιδιότητά μου αυτή και τώρα που τα γερμανικά μου τα εξάντλησα θα συνεχίσω στα αγγλικά. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Εργάζομαι για, μια, ε, για ένα πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα θέματα TBT και θα ήθελα να ομιλήσω και προσωπικά επί έξι χρόνια έχω εργαστεί και συνεργαστεί σε τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις και είναι μεγάλο το πάθος αυτής της εμπλοκής μου όμως προτού αναφερθώ σε κάποια από τα ξεχωριστά σημεία ας αναφέρω δύο επιφυλάξεις ως όρους η πρώτη επιφύλαξη. Είμαι οικονομολόγος για το θέματα εμπορίου. Αυτό είναι το αντικείμενό μου ως επιστήμονα και γνωρίζω ποια είναι η ισχύ του εμπορίου ως μέσο. Προσέρχομαι σε όλα αυτά τα θέματα του εμπορίου υπό αυτή την πτυχή, αλλά και έχοντας συνειδητοποιήσει ότι από μια χώρα και προερχόμενος είμαι και εξορισμού ένας ε, στην πρακτική εφαρμογή ε, συνεισφέρων στην ανάπτυξη μέσω του εμπορίου. Δεύτερον, γνωρίζοντας ότι αυτά τα θέματα αναφέρονται στις εμπορικές σχέσεις ΕΕ αφρικανικών χωρών, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση εγώ ίδιος προσωπικά να μην δώσουμε κάποια μαθήματα ή να κάνουμε κάποια κατήχηση τι θα πρέπει να κάνουν οι αφρικανικές χώρες και πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν. Θα έλεγα να είμαστε επιφυλακτικοί λοιπόν επ' αυτού. Αυτά που έχουμε κάνει. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για την ε, Καραϊβική. Τι γίνεται σε σχέση με αυτή την περιοχή του κόσμου. Απλά ποια μαθήματα μπορούμε να συναγάγουμε. Και να πω ότι πρώτα απ' όλα και κύρια πρόκειται για μια συμφωνία για την διακυβέρνηση διακυβέρνηση και διαχείριση θεμάτων εμπορίου. Κάποτε είπε κάποιος ότι οι συμφωνίες εμπορίου μοιάζουν, συγγενεύουν με τις ε, διατάξεις για τον αμοιβαίο αφοπλισμό. Συμφωνεί δηλαδή κάποιος να μην χρησιμοποιήσει, μην χρησιμοποιήσει κάποια μέσα πολιτικής, ιδιαίτερα εκείνα που θα μπορούσαν να ήταν βλαπτικά για την ε, ανάπτυξη για κάποιους άλλους. Υπό αυτό το πρίσμα ακριβώς ε, σε σχέση με αυτή την προσέγγιση έχουμε μια ομοιότητα με τον αφοπλισμό. Λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ισχύουν οι διατάξεις για τις επιδοτήσεις σε προϊόντα που έχουν συμφέροντα επ' αυτών οι χώρες της Καραϊβικής. Επίσης όλα αυτά κατοχυρώνονται και στην Συμφωνία Κοτονού θα θυμόσαστε ότι αυτές οι διατάξεις ε, για τις ε, διαπραγματεύσεις του τίτλου 2 σύμφωνα με, ε, με τη Συμφωνία του Κοτονού που είναι σαφής όσον αφορά τις αναφορές στα δικαιώματα του ανθρώπου. Όχι όμως μόνο στα δικαιώματα του ανθρώπου αλλά και στην χρηστή διακυβέρνηση. Και πάλι εδώ πρέπει να ενισχύσουμε και να ενδυναμώσουμε την παρατήρηση ότι αυτή η εμπορική συμφωνία αφορά την διακυβέρνηση και μάλιστα διακυβέρνηση και διαχείριση εμπορικών θεμάτων, αλλά κατοχυρώνεται και αγκυρώνεται όσον αφορά το ευρύτερο πλαίσιο της Συμφωνίας Κοτονού. Και εδώ έχουμε πολλά θέματα και αναφορές σε σχέση με αυτή τη συμφωνία, ξεκινώντας με το προήμιο ήδη και μια αναφορά στη Χάρτα των ε, Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου και μια αναφορά στη Σύμβαση και Προστασία των Θεμελιωδών Ελευθεριών και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την Χάρτα την Αφρικανική των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και στο άρθρο 1 της Συμφωνίας που πάλι ε, επαναλαμβάνει και κάνει λόγο για την ανάγκη να σεβόμαστε τα δικαιώματα των ατόμων το άρθρο 9 για τη δημοκρατία, τα δικαιώματα, τα δημοκρατικά και το κράτος δικαίου. Το άρθρο 2 για τον εκδημοκρατισμό, για την ανάπτυξη και την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Και το άρθρο 3 μετά στη συνέχεια που καθορίζει ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου αποτελούν τμήμα του πλαισίου χρηστής διακυβέρνησης. Αυτά όλα λοιπόν εντάσσονται στη Συμφωνία Κοτονού. Υπάρχουν όμως εξειδικευμένες ρυθμίσεις και πιο χειροπιαστά στοιχεία σε σχέση με την Καραϊβική και τη Συμφωνία για την Καραϊβική για τα δικαιώματα του ανθρώπου, πιο εξειδικευμένα. Προφανώς υπάρχει και η ανησυχία, το μέλημα ότι δηλαδή αν η Συμφωνία του Κοτονού και όταν εκπνεύσει το 2020 και συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε μια συμφωνία εμπορίου για την μεταγενέστερη περίοδο, τι θα γίνει σε σχέση με αυτά τα δικαιώματα του ανθρώπου ως τόξο μέσα, στα οποία, μέσα στο οποίο αυτό πλαίσιο είχαν τεθεί. Θα επιχειρηματολογούσα και θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη ΑΚΕ αντιμετωπίζουν τρεις προκλήσεις σε σχέση με την ανανέωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων. Ένα, το, η αναθεώρηση όσον αφορά τα θέματα status quo και αυτό πάλι αφορά την κατοχήρωση, ισχυρή κατοχήρωση των ε, δικαιωμάτων του ανθρώπου και της χρηστής διακυβέρνησης. Δεύτερον, η Συμφωνία Κοτονού θα επικαιροποιηθεί για να αντανακλά περισσότερο τις ε, διμερείς ε, διαπεριφερειακές σχέσεις. Δηλαδή, Αφρικανική Συμφωνία ΕΕ Αφρικανικών χωρών, συγκεκριμένες συμφωνίες όπου τα δικαιώματα αυτά κατοχυρώνονται από αμφότερες τις πλευρές, όχι μόνο στις ε, συμφωνίες εμπορίου, αλλά και στην συνεργασία για την ανάπτυξη και στα συγκεκριμένα πιο εξειδικευμένα μέσα και μέτρα και φυσικά στον πολιτικό διάλογο που ε, θα προάγεται. Και η τρίτη εναλλακτική επιλογή είναι η αναθεωρημένη επικαιροποιημένη συνθήκη Κοτονού, στην οποία θα διατηρηθούν οι τριυπηρωτικές ε, αυτές ρυθμίσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως η επικέντρωση θα είναι πιο αποτελεσματική στη λειτουργία. Δηλαδή, ώστε και οι δύο πλευρές να μπορούν να επιλέγουν με τέτοιο τρόπο το πλαίσιο, ώστε η χρηστή διακυβέρνηση να διασφαλίζεται από πλευράς πλαισίου. Υπό όλα αυτά θα έλεγα ότι σε σχέση με το μέλλον οι σχέσεις αυτές θα διαμορφωθούν σε σχέση με τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Τώρα, για τις διατάξεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου σε σχέση με αυτά, να πω το εξής. Βρίσκονται ήδη στο προήμιο. Είναι θεμελιώδη δικαιώματα μεγάλης εμβέλειας. Είναι μια πολύ σημαντική διάταξη μετά στο άρθρο 3 που αναφέρεται στην εφαρμογή αυτής της συμφωνίας λαμβάνοντας υπόψη είναι τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και δικαιωματικά όσον αφορά τους ανθρώπους ε, θέματα για τις μελλοντικέ γενναίες. Δηλαδή σε μια προσπάθεια συνολικά αηφόρου ανάπτυξης. Αλλά υπάρχουν και διατάξεις όσον αφορά τις αλλαδαπές άμεσες επενδύσεις όπου η συμφωνία για παράδειγμα επιτάσσει από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή να μην με περισταλούν περιβαλλοντικά δικαιώματα κοινωνικά δικαιώματα για να προσελκυστούν επενδύσεις. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική ε, παρατήρηση ως ε, ε, σχόλιο. Και εδώ σε σχέση με αυτό δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση που πίεσε να προαχθεί και να ενταχθεί αυτό το στοιχείο, αλλά εμείς από πλευρά ΣΑΚΕ και από πλευράς των θεσμικών διατάξεων και ρυθμίσεων εσείς ως Ευρωβουλευτές είμαι βέβαιος ότι θα γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα συμβουλευτικό σώμα που εμπλέκει τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους μια απόφαση του 2010 για το πώς δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η αντιπροσωπεία του θα εκπροσωπείται και μετά μια συμβουλευτική επιτροπή που θα προαγάγει το διάλογο σε σχέση με την κοινωνία των πολιτών και στη συνέχεια υπάρχει εν τέλει η αναθεώρηση και η εποπτεία. Ο καθηγητής Βάουτερς νομίζω αναφέρθηκε σε αυτό. Είναι μια ευκαιρία επειδή είναι μια νέα καινοτόμα συμφωνία για να εντείνουμε και να επικεντρωθούμε περισσότερο στην ανάπτυξη των βέλτιστων πρακτικών για το πώς αυτή η συμφωνία θα μπορεί να εποπτεύεται και να αναθεωρείται. Και τούτων λεχθέντων πρόεδρε να ολοκληρώσω λέγοντας να προτείνω ότι πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Ως προς τούτο, επειδή γνωρίζω από πρώτο χέρι ποια είναι η σπουδαιότητα των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην πρακτική εφαρμογή όλων αυτών, θα επιχειρηματολογούσα και θα έλεγα ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι πραγματικά εκείνη η πλατφόρμα που είναι η πιο ενδεδειγμένη για τα θέματα ανάπτυξη όμως να κρούσω κόδωνα κινδύνου εδώ αυτό να γίνει αναγκαίος επιτακτικός όρος και προϋπόθεση. Γιατί? Για τους εξής λόγους. Δεν θέλουμε αυτό να γίνει ένα μη δασμολογικό πρόσκομα ή εμπόδιο. Δεύτερος λόγος. Δεν επιθυμούμε, δεν θα θέλαμε να πληγούν τα κράτη και ιδιαίτερα τα αφρικανικά κράτη και να υποστούν επικρίσεις μέσα σε αυτό το πλαίσιο η αλλαγή δεν θα προέρθει χρησιμοποιώντας κάποιες επικρίσεις ε, ή καταγγελίες και κατηγορίες ε, με έναν ομό τρόπο. Θα πρέπει να, γίνεται, να γίνει αναφορά και σε ένα πρόσφατο άρθρο στην New York Times από έναν πραγματογνώμονα του Συμβουλίου της Ευρώπης που δείχνει ότι η ίδια η Ευρώπη έχει πάμπολες περιπτώσεις παραβιάσεων και παραβάσεων δικαιωμάτων του ανθρώπου. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί. Ολοκλήρωσα ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε και η συμπρόεδρος έχει τον λόγο. Ε, τώρα θα δώσω τον λόγο στον πρέσβη του Μαυρικίου που θα μας δώσει μία έτσι, θα μας κάνει μια παρουσίαση ε, για το τι συμβαίνει στην ε, νήσο αυτή. Μια και τα ξέρει από κοντά. Και το πώς αναπτύσσονται, θα μας μιλήσει για το πώς αναπτύσσονται τα, πώς εξελίσσονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και πώς επηρεάζονται από τις συμφωνίες αυτές στην περιοχή του. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και Αντιπρόεδρε. Ο Πρόεδρος είπε ότι είμαστε εμπειρογνώμονες στον κλάδο σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ τον εαυτό μου εμπειρογνώμονα. Ε, είμαι από μια χώρα η οποία έχει αποδείξει ότι πιστεύει στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου. Είμαι εκπρόσωπος του Μαυρικίου, μιας χώρας που εφαρμόζει μια προσωρινή Συμφωνία Οικονομική Εταιρική Σχέση μαζί με κάποιε άλλε χώρε τη Αφρικανική Υπήρου. Και είμαστε η πρώτη περιοχή τη Αφρική που εφαρμόσουμε μια τέτοια Συμφωνία Εταιρική Σχέση. Δεν πρόκειται λοιπόν να σα δώσω μια πλήρη εικόνα τη Αφρική για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά ελπίζω να μπω σε κάποια από τα θέματα, τα οποία είναι σημαντικά για την Αφρική πάντως. Ο κύριος Λότζος, συνάδελφός μου, ξεκίνησε την συζήτηση εγώ δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειε. Ε, μίλησα για τη τρέχουσα κατάσταση, όπου στη Συμφωνία Κοτονού έχουμε διάφορα άρθρα τα οποία μιλάνε για τον πολιτικό διάλογο, για τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Αναφέρθηκε στο άρθρο 8-9, 96-97 που είναι σημαντικά για τα θέματα αυτά σημαντικά θα της Συμφωνίας Κοτονού. Η συμφωνία αυτή είναι μια συμφωνία πλαίσιο, η οποία έχει συμβατικέ υποχρεώσεις, ε, επιβάλλει συμβατικέ υποχρεώσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στι στις χώρες ΑΚΕ. Επίσης είναι και ένα αναπτυξιακό εργαλείο, ένα πλαίσιο που επιτρέπει όχι μόνο το εμπόριο, αλλά και την βοήθεια, την αναπτυξιακή βοήθεια σε κάποιο βαθμό. Είναι δυνατόν λοιπόν σε τέτοιου τύπου συμφωνίες να υπάρχουν στοιχεία τα οποία μας αναγκάζουν να προωθήσουμε το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη χρηστή διακυβέρνηση κτλ. Τώρα πλησιάζουμε όμως ε, στο τέλος συμφωνίας Κοτονού, δηλαδή το 2020, λίγη συμφωνία αυτή και δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Και αν ο τίτλος 2 της συμφωνίας Κοτονού δεν ισχύει πια και θα πρέπει να διαπραγματευτούμε τέτοιες συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, μπορεί να προβληματιστούμε με έναν τελείως καινοτόμο τρόπο. Πολλές από τις εμπορικές προτιμήσεις που υπάρχουν, που υπήρχαν τις παλιές μέρες, τα Starbucks, το πρωτόκολλο της ζάχαρης, όλα αυτά τέλειωσαν. Και μπαίνουμε σε αυτές τις νέες εμπορικές ε, διευθετήσεις. Επίσης, η γεωπολιτική κατάσταση στο μεταξύ έχει αλλάξει. Όπως είπε και η Επίτροπος Μάλστρομ της προάλλες, ήταν σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαπραγματευτεί τη συμφωνία TTIP. Γιατί η δύναμη της φωνής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώνεται. Και στην Αφρική επίσης πρέπει να υπάρξει προσοχή γιατί υπάρχει, υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί εταίροι οι οποίοι δρούν, παίζουν στην Αφρικανική Ήπειρο και κάνουν πολλά πράγματα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν προσέξει πολύ, μπορεί να χάσει αυτό το παγκόσμιο ρόλο που έχει στην Αφρική. Επίσης υπάρχει μια μεγαλύτερη αφύπνιση των Αφρικανών και της, ε, του δυναμικού που έχει η Αφρική, τους, αφύπνιση για τους πόρους που έχει η Αφρική και αυτό θα πρέπει ε, να ληφθεί υπόψη. Και δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν παλιά. Και γι' αυτό οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ε, μας πήραν τόσο καιρό για να συναυθούν. Και δεν ξέρουμε αν σε όλες ε, τις περιπτώσεις θα έχουμε μια τέτοια συμφωνία σε αυτό το νέο πλαίσιο λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Αντιπρόεδρος είπε κάτι πολύ σημαντικό, μια σημαντική φράση. Είπε ότι θα πρέπει να υπρασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός και εκτός των συνόλων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα πρέπει να γίνει με έξυπνο τρόπο. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εκεί ακριβώς ε, θα πρέπει να εστιάσει όλη η συζήτηση. Ποιο είναι αυτός ο έξυπνο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για την Αφρική, καταρχά, όταν μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για θεμελιώδη δικαιώματα, να μην ξεχνάμε ότι το δικαίωμα στην ανάπτυξη θεωρείται επίση σημαντικό και θεμελιώδη δικαίωμα. Επομένω, όπω είπε και ο κύριος Λότζ, όταν μιλάμε για το εμπόριο, θα πρέπει να εξετάζουμε το εμπόριο από αναπτυξιακή σκοπιά. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το εμπόριο γίνεται ατμομηχανή ανάπτυξης ατμομηχανή εσόδων, εισοδημάτων, απασχόλησης και άρα εξάλληψης της Θα πρέπει λοιπόν αυτό να ληφθεί υπόψη. Όταν μιλάμε για τις κυρώσεις, όταν μιλάμε για μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν, μιλάμε για την εκτέλεση, για τις ρήτρε μάλλον εκτέλεσης. Μην ξεχνάμε ότι αυτό θα είναι στο πιο δύσκολο πράγμα να κάνουμε. Δηλαδή στην Αφρική και σε διάφορες αφρικανικές περιοχές κινούμαστε προς την ολοκλήρωση, προς την ενοποίηση, προς μια ενιαία τελωνιακή, έναν ενιαίο τελωνιακό χώρο, μια τελωνιακή ένωση. Αν επιβληθούν κυρώσεις σε μια χώρα, τότε πρέπει να δούμε αν μπορούμε να επιτρέψουμε σε όλες τις χώρες της περιοχής να υποφέρουν, γιατί δεν γίνεται να επιβάλλεται κυρώσεις εναντίον μίας μόνο χώρα όταν όλες αυτές οι χώρες δημιουργούν, αποτελούν μία τελωνιακή επικράτεια. Επομένως, τι μπορεί να γίνει. Πιστεύουμε ότι στην Αφρικανική Ήπειρο υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν προωθηθεί. Έχουμε τον ΕΠΑΤ, το Μηχανισμό Ισότιμης Αναθεώρησης της Αφρικής, Peer Review Mechanism, και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεργαστεί με αυτές τις οργανώσεις και να δει πώς θα μπορούσε να συζητήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ε, είτε από περιφερειακή σκοπιά είτε από υπηρετική σκοπιά ε, πάντω με συλλογικό τρόπο. Δεν ξέρω πώ μπορεί να γίνει. Αν γίνει τιμερό μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και μία επιμέρου ε, χώρα, θα υπάρξουν τεράστια θέματα. Πρόσφατα έγινε μεγάλη συζήτηση για την ε, ομοφιλοφιλία, α πούμε, στην Αφρική. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτά τα θέματα, παρότι είναι τώρα πολύ σημαντικά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνές επίπεδο στην Αφρική, είναι πάντα, παραμένουν πολιτιστικά θέματα και σε πολλές περιπτώσεις, όπως είδαμε και στο παρελθόν, οι νόμοι που ισχύουν για θέματα, ας πούμε, ομοφιλοφιλίας, είναι νόμοι οι οποίοι έχουν επιβληθεί από τους απεικιοκράτες και δεν έχουν αναθεωρηθεί ποτέ. Τι οι νόμοι που τους έφεραν οι απεικιοκράτες πρέπει να μας λένε οι ίδιοι απεικιοκράτες, οι πρώην απεικιοκράτες τέλο πάντων, ότι πρέπει να τους α, να τους ακυρώσουμε. Υπάρχει κάτι το σημαντικό εδώ, η μεταρρύθμιση βέβαια. But you have to give time. Πρέπει να τους κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις, αλλά πρέπει να δώσουμε χρόνο για να γίνουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις. move. Ο καλός τρόπος είναι να περάσουμε στο, από το σύστημα που έχουμε τώρα, όπου εφαρμόζουμε κυρώσεις, ε, σε ένα σύστημα που θα συνεργαστούμε συλλογικά με τις ε, αφρικανικές περιοχές και με την Αφρικανική Ένωση για να μπορέσουμε να εξετάσουμε από κοινού τα προβλήματα. Αυτά είναι κάποια από τα στοιχεία που θα ήθελα να σας ε, υπογραμμίσω. Και εμείς ευχαριστούμε πρέσβη. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ζακ Μπερτελό, που είναι οικονομολόγος ε, για, τη Γεωργία, ε, δουλεύει στην ε, ΜΚΟ Αλληλεγγύη με έδρα την Τουλούζη. Και ξέρει πάρα πολύ καλά, έχει μεγάλη εμπειρία για θέματα Δυτικής Αφρικής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεδομένου του περιορισμένου χρόνου θα εστιαστώ στη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με τη Δυτική Αφρική και δεν αμφισβητώ την αρισιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία αποτελεί κομμάτι όλων των εμπορικών συμφωνιών εδώ και 30 χρόνια αλλά ποτέ δεν τηρήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έδωσε το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων στο Πακιστάν ε, που έχει το ρεκόρ του κόσμου για τις παρεμβάσει των δικαιωμάτων των γυναικών και των δολοφονιών ατόμων και δεν ελήφθη υπόψη ούτε για τη συμφωνία με την Κεντρική Αμερική ούτε για τη συμφωνία με την Κολομβία όπου έχουμε παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις παραστηριωτικές οργανώσεις. Ε, δέκα χώρες έχουν εξαιρεθεί Ερυθρέα, Σουδάν, Κονγκό κτλ. Αυτή η νέα συμφωνία ανταποκρίνεται σε άνηση μεταχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπογράφει ε, μη ισορροπημένες ε, εμπορικές συμφωνίες που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι οι συμφωνίες αυτές ε, ε, ήδη υποβαθμίζουν τις οικονομικές δυνατότητες των χωρών αυτών, ε, την ε, πρόσβαση σε τρόφιμα και με διάφορες άλλες επιπτώσεις, ενώ συνεχίζουν να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Χωρίς αυτές τις συμφωνίες η Αφρική έχει να αντιμετωπίσει την υπερθέρμανση του κλίματος και τα δημογραφικά προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα πρώτη, πρώτα απ' όλα η απώλεια των ε, τελωνιακών τελών θα ήταν τεράστια για την Ιγυρία ε, βάσει στοιχείο της Παγκόσμιας Τράπεζας ε, είναι λανθασμένη. Δεν είναι σοβαρά τα στοιχεία που δίνονται επί 20 ετών. Ο πληθυσμός της Δυτικής Αφρικής μέχρι το 35 θα αυξηθεί κατά 67% θα είναι ίσο πληθυσμό τη Δυτική Αφρικής μέχρι το 2031 με τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Παγκόσμια Τράπεζα δεν υπολογίζει την απώλεια τελών και την απώλεια ΦΠΑ κατά την εισαγωγή. Το South Center έχει ξανακάνει τους υπολογισμούς και η Solidarité τους έχει συμπληρώσει βάσει του 2014 τα ετήσιες ζημίες ε, το 2020 θα ανέλθει από 1,4 δισεκατομμύρια σε πολύ περισσότερο το 2035. Δεδομένων αυτών των τεράστιων ζημιών, οι αντιστοιχνιστικές βοήθειες που προβλέπονται στο άρθρο 60 ε, δεν είναι ρεαλιστικές. Η DG Τεύκο επιβεβαίωσε τον Ιούνιο ότι δεν μπορεί να δοθεί επιπλέον βοηθεία για τέτοιε συμφωνίε. Αντισταθμίζονται αυτέ οι απολύσει με άνοδο τη φορολογία εσωτερικά στι χώρε, αφαιρώντα ε, ε, χρήματα από την εκπαίδευση και τη γεωργία και να μην μιλήσω για τη Συμφωνία Διευκόλυνση των Συναλλαγών. Deuxième η μελέτη για την Ιγυρία της Παγκόσμιας Τράπεζας το 2014 προβλέπει άνοδο μεγάλη των κερδών των καταναλωτών, αλλά αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Θα βασιστεί στη μείωση των τιμών των εισαγόμενων προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω των διατροφικών, το οποίο θα μειώσει την τιμή των τοπικών δημητριακών, τον, του γάλακτος και θα φτωχύνει τους γεωργούς που αποτελούν το 61% του ενεργού πληθυσμού διότι αντίθετα από ό,τι υπόθηκε το 23 Ιουνίου είπαν η κυρία Γκαλέ και ο το 35% των τροφίμων δεν εξαιρούνται από την απελευθέρωση τα δημητριακά, το ρύζι και το γαλασκόνι Το 69% λοιπόν των Ιγυριανών ζουν κάτω από το κατόφλιο της φτώχειας, του 1 δολαρίου την ημέρα. Και εδώ επανέρχομαι στα όσα υπόθηκαν προηγουμένως, οι εξαγωγές δημητριακών έλαβαν το 13 τεράστιες επιδοτήσεις. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι δεν επιδοτεί τις εξαγωγές, αλλά ξεχνά ότι τέσσερις φορές στον ΠΟΕ κρίθηκε ότι οι εσωτερικές επιδοτήσει ε, στο εξαγόμενα προϊόντα αποτελούν κομμάτι του Η κυρία Γκαλίνα επίση δεν ανέφερε την έκθεση που παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Απριλίου του 2014 βάσει κειμένου τη ε, συμφωνία, που έχει πολύ αρνητικά συμπεράσματα. Άνοδο της ανεργίας, μείωση του προπολογισμού και μείωση του ΑΕΠ. Και όλα αυτά έγιναν πριν από την κατάρρευση των τιμών του πετρελαίου και το IMF προβλέπει μείωση των πετρελαϊκών εσόδων της Νιγηρίας το 2015 που θα μειώσει τις δημόσιες επενδύσεις και την ανάπτυξη. Η μείωση των εσόδων σε συνδυασμό με την ανάγκη καταπολέμησης της Μποκοχαράμ που έτσι στρατολογεί ακόμη πιο εύκολα τον κόσμο με την ανατολή στόχιας οδηγεί σε μείωση των δαπανών υγείας και εκπαίδευσης. Τρίτη αιτία, οι κανόνες του ΠΟΕ ε, σέβονται πολύ περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε διαμαρτυρίες από τις χώρες του EPC. Ε Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεχόμενη να μειώσει τα τελεινικά τέλη για τις αγωγές μπανάνας με τις διμερείς συμφωνίες ε, του 2012 με την Κεντρική Αμερική, την Κολομβία, το Περού και τον Ισημερινό το 2014. Έτσι αυτές οι χώρες δεν έχουν πλέον ένσταση για επιστροφή στις εμπορικές προτιμήσεις του ΛΟΜΕ. Και μάλιστα υπήρξε και εξαίρεση για τη Μολδαβία το 2008. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να υποστηρίξει το αίτημα της ε, Αφρικανικής Ένωσης να αναγνωριστεί η περιοχή ως μεγάλη ε, περιοχή PMA, διότι όλες αυτές οι χώρες ε, πληρούν τα κριτήρια. Η απέτηση μείωση των τελωνικών τελών κατά 80% έρχεται σε αντίθεση με την αρχή όλα εκτός όπλων, αλλά και με όλες τις συμφωνίες του ΠΟΕ που δεν απαιτούν εμπορική αμεβαιότητα για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Δηλαδή αντί να τα μειώσουμε κατά 80% θα μπορούσαμε να ε, χαμηλώσουμε κατά πολύ μικρότερο ποσοστό. Οι χώρες απεσέ επίσης δεν πρέπει να συνάπτουν τις συμφωνίες αυτές Ε, το 2008 προβλέφθηκαν ρήτρες ε, διασφάλισης ε, καλύτερες από τις Ευρωπαϊκές Συμφωνίες και σύμφωνα με το ΦΑΟ η τοπική οικονομική κοινότητα γίνεται μέλος του ΠΟΕ για παγιωμένα δικαιώματα. Τέλος, οι πολλές διμερείς συμφωνίες, TTIP για παράδειγμα και η ΣΕΤΑ θα οδηγήσουν σε αύξηση των εμπορικών ε, σόδων. Γιατί λοιπόν ε, επιβάλλουμε τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης λόγω της πίεσης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στα κράτη της Δυτικής Αφρικής. Ε, πίεσης μεγάλων ομίλων, γαλλικών μάλιστα, η εταιρεία φρούτων που εξάγει τις περισσότερες μπανάνες και δωρονά από την Κάνα και το ακτή ελεφαντοστού άσκησε πίεση για, πίεση για να μην πληρώσει τα σχετικά τέλη. Ο όμιλος Νιμράν από τον Τακάρ και τον Αμπετσάν πέτυχε μείωση των τελών για τα Δημητριακά και το ρύζι. Και ο όμιλος Μπολορέ που ασχολείται με όλες τις λιμενικές εγκαταστάσεις του κόλπου της Γουινέας συμμετέχει στην εξαγωγή των δύο τρίτων του κακάο από την ακτή ελεφαντοστού. Μιλάμε για 164 ε, ε, εκατομμύρια ευρώ τελών που θα χαθούν εάν τεθεί σε ισχύ η συμφωνία. Αλλά τα τέλη που καταβάλλονται ε, αντιστοιχούν στο 4,4% απώλειας τελωνιακών εσόδων ε, της Δυτικής Αφρικής το 2050 και το 6% το 2035 εφόσον εφαρμοστεί η συμφωνία. Γι' αυτό το λόγο η κοινωνία των πολιτών της Δυτικής Αφρικής ζήτησε το 16 κράτη να συνεργαστούν ε, για να πληρώσουν εξαγωγή των χωρών αυτών τα 164 εκατομμύρια που αντιστοιχούν όπως είπα το 6% των, μόνο των ζημιών. Ε, θα σήμαινε αυτό συμμετοχή ε, επιδότηση 2,2% των εξαγωγών τους. Merci Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα έχετε εσείς τον λόγο παρακαλώ, Λουτ. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ τους τέσσερις ε, προλαλήσαντες πραγματογνώμονες. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση των τεσσάρων αυτών προσεγγίσεων. Και όσον αφορά τη Συμφωνία για τις χώρες της Δυτικής Αφρικής, βλέπουμε ότι πολλά από τα σημεία που αναφέρθηκαν για τη συζήτηση, την ευρύτερη συζήτηση όπως τίθενται καθώς συνεχίζουμε. Θα ήθελα να επανέλθω στα θέματα συγκεκριμένα των ρητρών για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Έχω κάποιες σύντομες ερωτήσεις που στοχεύουν συγκεκριμένους ε, πραγματονόμονες. Τον κύριο Βάουτες, υπό το δικό σας πρίσμα, πώς νομίζετε ότι μπορούν οι όροι και προϋποθέσεις ε, του, της Συμφωνίας Κοτονού όπως εντάσσονται σε αυτές τις συμφωνίες να λειτουργήσουν σε ένα νομικό πλαίσιο. Αυτό το πλαίσιο για τα δικαιώματα του ανθρώπου σε σχέση με τις αρχές του Κοτονού θα μπορούσε να επιβιώσει σε όλα τα πλαίσια που αναφέρονται και από τον κύριο Λότζ για το τι θα συνέβαινε μετά τη Συμφωνία Κοτονού, την εκπνοή της. Ποιες επιπτώσει θα υπήρχαν αν υπήρχε μια νέα Συμφωνία Κοτονού ή αν εξέπνε η Συμφωνία Κοτονού. Προ τον κύριο Λότζ, την παρέμβασή σα την βρήκα πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα θα ήθελα να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στην, στα βιώματα των καραϊβικών χωρών. Επί τρία χρόνια έχουμε το θέμα της εφαρμογής ε, αυτών των ε, πλαισίων. Είναι διαφορετικά από τις συμφωνίες ε, για τις χώρες της Αφρικής θεσμικά. Έχουμε ένα κεφάλαιο που αφορά την αηφόρο ανάπτυξη, έχουμε τα θεσμικά όργανα και τον διάλογο επιπλέον Αναφερθήκατε σε αυτά στο τέλος της παρεμβασής σας. Θα έλεγα αυτό που είπατε για το ότι η αλλαγή προέρχεται από την εμπλοκή σε αυτό το έργο είναι ακριβώς οι επικρίσεις που ασκούμε εμείς, ή τουλάχιστον εγώ προσωπικά, σε κάποιες από τις αφρικανικές αυτές συμφωνίες, όπου δεν υπάρχει η συμμετοχή της ε, ε, κοινωνίας των πολιτών, ε, όπως σε άλλα πλαίσια. Με ενδιαφέρει λοιπόν να ακούσω για την Καραϊβική τι γίνεται σε σχέση με την συμφωνία αυτή για την εποπτεία, ιδιαίτερα το κεφάλαιο 5, κοινωνικές περιβαλλοντικές πτυχές και τα δικαιώματα τα εργασιακά που εμπίπτουν και στα δικαιώματα του ανθρώπου μια και είναι άρρηκτα και δεν μπορούν να τεμαχιστούν και είναι οικουμενικού χαρακτήρα και πώς ε, υπάρχει, πώς διαμορφώνεται η εργασία καθημερινά από πλευρά τη Επιτροπή. Είναι ο σωστότερος τρόπο εποπτείας. Με ενδιαφέρει πολύ η άποψή σα. Στη συνέχεια, η τελευταία μου ερώτηση θα ήταν, μια και ακούσαμε πολλές από τις επικρίσεις, ίσως θα το προφέρω λάθος το όνομα, του κυρίου Μπερτελό για τις επικρίσεις που έχουν ασκηθεί. Θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι το ιδανικό πλαίσιο σύμφωνα με την άποψή σας για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα του ανθρώπου και να επιβληθεί ο σεβασμός ε, της εφαρμογής των δικαιωμάτων αυτών. Τι θα έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα μπορούσαν οι περιφερειακές αυτές συμφωνίες να χρησιμοποιηθούν για να συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση. Επανέρχομαι σε ένα σημείο από τους προλαλήσαντες, από τον πρέσβη του Μαυρικίου και τον κύριο Λότζ, ότι το εμπόριο είναι το κλειδί για την ε, για το θεματολόγιο, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για την ανάπτυξη. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι συμφωνίες εμπορίου θα είναι φορείς και οχήματα για αυτή την ανάπτυξη και την προαγωγή στην ανάπτυξη και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Βερζιά παρακαλώ. Euh, euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για όλες τις παρουσιάσεις. Ήθελα απλά να επισημάνω στους δύο προεδρούς ε, ότι εδώ υπάρχει ο Μαμαντού Σισικό και από τη Σενεγάλη, πρόεδρος του δικτύου των ε, χωριών και Επενδιοργών, ε, μέλος της πλατφόρμας των Αφρικανών χωρικών και πιστεύω ότι θα έπρεπε να ακούσουμε την άποψή του για τα ζητήματα δικαιωμάτων και οικονομικής ανάπτυξης των Αφρικανικών χωρών. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω λοιπόν να ακούσουμε και αυτό τον κύριο. Έχω τρεις ερωτήσεις, πιο συγκεκριμένες. Η πρώτη, αναφερόμαστε σε αυτή τη ρήτρα δικαιωμάτων, ανθρώπινων δικαιωμάτων συνέχεια και βιώσιμης ανάπτυξης. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτές τις δύο έννοιες σε μια συμφωνία και ταυτόχρονα να βάζουμε σε αυτές τις συνθήκες, όπως βλέπουμε στις συμφωνίες ε, να έχουμε μηχανισμούς που υπονομεύουν το ζήτημα των δικαιωμάτων. Ε, και το είδα προηγουμένως όταν συζητούσαμε για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων ή την ελευθερία του τύπου ή το δικαίωμα για δημοκρατική οργάνωση των εκλογών. Ξέρετε, αλλά υπάρχουν και όλα τα παράγωγα δικαιώματα ε, της ανάπτυξη, για παράδειγμα το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Ε, στην έχουμε περιπτώσεις αρπαγής γεών στην Αφρική. Πώ οι συμφωνίε αυτέ που διαπραγματευόμαστε τώρα εμποδίζουν το μονοπόλιο της γης από μια οικονομική ανάπτυξη που δεν ε, είναι εποφελής για τους τοπικούς πληθυσμούς. Το δικαίωμα για την ε, ε, διατροφική κυριαρχία, όχι την ασφάλεια, δηλαδή κάθε χώρα να έχει τη δυνατότητα να καλύπτει τις ανάγκες του πληθυσμού αλλά έχουμε και μηχανισμούς που τροφοδοτούν σειράξεις υπάρχουν δομικοί μηχανισμοί που ε, τροφοδοτούν σειράξεις σε αυτές τις χώρες, ε, μέσα σε αυτές τις συμφωνίες. Πώς μπορούμε λοιπόν να έχουμε συνεκτικές πολιτικές. Ρώτησα χθε την Επιτροπό μάλιστα αλλά δεν έλαβα απάντηση δυστυχώς. Ίσως να λάβω κάποια απάντηση σήμερα από τους ομιλητές μας. Ποια θα ήταν η καλύτερη δυνατή συμφώνια που θα επέτρεπε να έχουμε συνοχή πολιτικών. Κατά την απόψή μου και το είπατε, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι το αποτέλεσμα της ρεσιμότητας. Αντιθέτως, είναι το αποτέλεσμα των όσων θα μπορέσουμε να κάνουμε με συνοχή με εσά για αυτέ τι χώρε. Το δεύτερο ερώτημα είναι ο ρόλο τη κοινωνία των πολιτών. Γνωρίζουμε δύσκολη είναι η διαπραγμάτευση τέτοιων εμπορικών συμφωνιών. Το βλέπουμε και εδώ στην Ευρώπη. Το ζήτημα τη μη διαφάνεια αυτών των διαπραγματεύσεων. Ξέρουμε ότι η κοινωνία των πολιτών στην Αφρική δυσκολεύεται με αυτέ τι διαπραγματεύσει δυσκολεύεται να συμμετάσχει. Πώ μπορούμε να την κάνουμε να συμμετάσχει την κοινωνία των πολιτών τη Αφρική και τη Ευρώπη, ώστε να διατυπώνουμε καλύτερα αυτέ τι συμφωνίε, να τι συντάσσουμε καλύτερα, ώστε να υπάρχουν κάποιε μελέτε επιπτώσεων εκ των προτέρων που θα λαμβάνονται υπόψη. Πραγματικά όμω, γιατί άκουσα ότι η Κομισιόν δεν έλαβε υπόψη ορισμένε μελέτε που ε, καταδείκνυαν αποτελέσματα όχι πολύ θετικά σε σχέση με αυτά που θεωρούσαμε εμεί ότι υπάρχουν. Πώ λαμβάνονται λοιπόν, πώ μπορούν να λαμβάνονται υπόψη τέτοιε μελέτε και να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών. Και τέλος αναφέρεται ότι οι, Ευρω... οι επικρίνουν ιδιαίτερα τον τρόπο διαπραγμάτευσης των ε, συμφωνιών αυτών από την Ευρώπη. Δηλαδή οι ΗΠΑ σέβονται καλύτερα ε, την Αφρική. Με ποιο τρόπο, τι μοντέλο χρησιμοποιούν, ε, πώς θα μπορούσε αυτό να μας εμπνεύσει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστούμε πολύ, David Martin. Ευχαριστώ, Πρόεδρε ως μέλος και των δύο επιτροπών για τα δικαιώματα του ανθρώπου και της Επιτροπής Εμπορίου το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα και θέλω να ευχαριστήσω τους τέσσερις πραγματογνώμονες που θεωρώ ότι οι εισηγήσεις τους ήταν πάρα πολύ επικοδομητικές. Αλλά περισσότερα ερωτήματα τίθενται από ότι δίνονται απαντήσεις. Και η γενική αυτή παρατήρηση σε σχέση με τον καθηγητή Βάουθες που είπε ότι δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο για τα δικαιώματα του ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις συμφωνίες εμπορίου, αλλά διαφοροποιούμαστε. Έχουμε όλοι κάποιες ιδέες γιατί συμβαίνει αυτό και διαφοροποιούμαστε στο επιστημονικό επίπεδο. Γιατί, λόγω της οικονομικής αντιμετώπισης εκείνων με τους οποίους διαπραγματευόμαστε, λόγω κάποιων διασυνδέσεων, επειδή εμπιστευόμαστε κάποιες χώρες περισσότερο από κάποιες άλλες, ε, λόγω του ότι για παράδειγμα υπάρχουν αυτές οι διαφορές ε, που δημιουργούν ε, αυτό το πλαίσιο. Και πιο συνδεδεμένο με το σημερινό θέμα <clears throat> είναι σε σχέση με την Cariform για τις χώρες της Καραϊβικής ένα θετικό πλαίσιο όσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου, τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά δικαιώματα και ακούμε από πλευρά της ε, Επιτροπής τα σχετικά, εγώ μας γνωρίζω και θα έλεγα ότι όταν πήγε να διαπραγματευτεί με τις ε, χώρες της Αφρικής ε, η Επιτροπή, δεν υπήρχε η ικανότητα να επιτευχθεί αυτό. Διερωτώ με, γιατί ήταν οι χώρες της Αφρικής, είχαν περισσότερες αντιστάσεις σε σχέση με την προσέγγιση των χωρών της Καραϊβικής στο Κάρινφορν. Και στη συνέχεια αναφέρθηκε ένα πολύ σημαντικό θέμα αναλώνουμε πολύ χρόνο συζητώντας αυτά τα θέματα και το περιεχόμενο των διατάξεων και ρητρών για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Τώρα πρέπει να δούμε την επίπτωση σε σχέση με το αποτέλεσμα και να δούμε ε, ε, το ότι θα μπορούσαμε να είχαμε ίσως καλύτερα αποτελέσματα. Θα ήθελα να μου πείτε θα ήταν διαφορετικά τα αποτελέσματα αν υπήρχε διαφοροποιημένη προσέγγιση σε σχέση με αυτές τις συμφωνίες εμπορίου. Δεν είμαι προκατηλημένος, αλλά η ύπαρξη των μη, ε, της μη εκτέλεσης, κάποιων ρητρών μη εκτέλεσης, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιούμε, ίσως ε, θα μπορούσαν ε, να έδιναν κάποια επιχειρήματα. Δεν ξέρω, συμβαίνει αυτό, είναι η πραγματικότητα ή όχι. Και εν τέλει πολλές άλλες ερωτήσεις, αλλά πρέπει να σταματήσω σε αυτό το σημείο και να επανέλθω σε σχέση με το current form για τις χώρες της Καραϊβικής. Η δική μου στα, σε μισό λεπτό αντιμετώπιση με τα βιώματά μου είναι ότι είναι εξαιρετικό αυτό το πλαίσιο της συμφωνίας αλλά τα αποτελέσματα ήταν πενιχρά, ήταν γλίσχρα. Κατά τα τελευταία χρόνια μόνο μία ουσιώδη συνάντηση είχαμε στην Καραϊβική με τους εταίρους ε, των χωρών αυτών και μία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έγινε σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο. Η παρακολούθηση λοιπόν, η συνέχεια που δόθηκε κοινοβουλευτικά δεν ήταν θετική όπως θα έπρεπε και θα πρέπει ίσως να δούμε μια βελτίωση των πραγμάτων και να πάρουμε στα σοβαρά το τι μπορεί να γίνει. Δεν είναι θέμα μόνο να ενταχθούν στις συμφωνίες αυτές οι ρήτρε, αλλά να υπάρχει και η συνέχεια. Ευχαριστώ. Πολύ σωστά τα λέτε, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Παντσέρη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Το 2014 στην Αφρική υπήρξε καταστρεπτικό έτος για την υπερασπίση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Όσοι τα υπερασπίζονταν βρέθηκαν παγιδευμένοι σε εμπόλεμες περιοχές. Οι κυβερνήσεις στα λόγια υποστηρίζουν την προστασία των πολιτών, αλλά οι τάξεις των κυριάρχων στον κόσμο τους πρόδωσαν αυτή είναι η εισαγωγή της ετήσιας έκθεσης 2014-2015 ε, της Amnesty International, της Διεθνούς Αμνηστίας. Η κατάσταση είναι αυτή. Παρότι εμείς ε, συχνά στρέφουμε τα ματιά αλλού και πώς πρέπει να το δούμε όλο αυτό. Ευχαριστώ φυσικά τους εμπειρογνώμονες ε, που ήρθαν εδώ σήμερα το πρωί, αλλά πρέπει να πω και θέλω να το συζητήσουμε μαζί. Μου φαίνεται ότι συχνά εύκολα μπορεί να δει κάποιο δύο προβλήματα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικότερα στην Αφρικανική Ήπειρο. Πρώτον, το θέμα της realpolitik, της ε, πραγματική πολιτικής. Δεν μπορούμε να ε, λέμε ότι βάζουμε όλες αυτές τις ρήτρε και τι βάζουμε σε τόσο μεγάλο βαθμό γιατί έχουμε ένα μεγάλο ανταγωνιστή την Κίνα η οποία Κίνα εφαρμόζει τις ε, πολιτικές ε, υποδομών και όλα αυτά χωρίς τέτοια δικαιώματα. Οπότε και εμείς με κάποιο τρόπο πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό. Αυτό είναι το πρώτο θέμα ε, συζήτησης που πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή. Το δεύτερο σημείο, το άκουσα και σήμερα από τον πρέσβη του Μαυρικίου, είναι ότι χρειάζεται χρόνος. Πόσος. Πόσος χρόνος. Εντάξει, έχουμε τις παραδόσεις, ε, έχουμε τις απεικιοκρατικές παραδόσεις κτλ. Ε, τρία υποθετικά σενάρια εργασίας ε, πιστεύω που θα πρέπει να σκεφτούν οι εμπειρογνωμονές μας. Πρώτα απ' όλα έχουμε τη Συμφωνία της Κοτονού. Είχαμε δύο αναθεωρήσεις τα τελευταία χρόνια. Την αναθεώρηση του 2005, την αναγνώριση του 2005 του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου το 2010 είχαμε μια δεύτερη αναθεώρηση η οποία ακόμα βρίσκεται σε φάση επικύρωση. Το 2013 την επικύρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πολλές επιφυλάξεις για διάφορα σημεία της συμφωνίας που δεν αποτυπώνουν τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ειδικότερα όσον αφορά τις αξίες. Για παράδειγμα, ατέθηκε το θέμα διακριτική μεταχείριση μεταχείρισης ε, ατόμων διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού. Δεν προβλέπεται καμία αναθεώρηση για το 2015 και εμείς αντικειμενικά θα μπορούσαμε να απαιτήσουμε στο 2015 να γίνει αναθεώρηση αυτής της συμφωνίας διότι χρειαζόμαστε μια βαθιά επικαιροποίηση της ε, συμφωνίας του Κοτονού. Το δεύτερο σημείο αφορά την αρισιμότητα. Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να εισάγουμε πιο αυστηρούς κανόνες αρισιμότητας ε, ώστε να ξεκινήσει συζήτηση, κάποιοι προβληματισμοί και να υπάρξει και μια θετική σχέση με την κοινωνία των πολιτών για να υλοποιηθούν οι στόχοι αυτοί. Το τρίτο σημείο, για να βγούμε λίγο και από τα καθαρά θεωρητικά ερωτήματα, για ποιο λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ζητά να ξεκινήσει ένα επίσημο φόρουμ για παραδείγμα στο πλαίσιο των διαφόρων συζητήσεων περί διεθνούς εμπορίου και αυτό το φόρμα αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος ε, για να ερμηνεύσουμε τις προσδοκίες και τις απαιτήσει ε, της αφρικανικής κοινωνίας ε, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Σατζεντίνη. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δυσκολεύομαι λίγο με τον ορισμό. Κάποιες δυσκολίες έχω με τους ορισμούς για τα πράγματα τα οποία συζητάμε. Για παράδειγμα, δώσατε το παράδειγμα των κόκκων κακάο από τη Δυτική Αφρική που οι συγκομιδές ε, καλύπτουν με παιδική εργασία, κάτι το οποίο δεν θέλουμε με κανένα τρόπο να γίνεται. Και το παράδειγμα του πρέσβη και τους ε, νόμους που θεσπίστηκαν από την απεικιοκρατία θα έλεγα είχαμε και εμείς αυτή την νομοθεσία αλλά την αλλάξαμε. Θα μπορούσατε και εσείς αλλά όμως εδώ είναι μια σαφής περίπτωση αυτή. Άλλα παραδείγματα μπορούν να δείξουν πως δεν θα θέλαμε να έχουμε εμπορικές σχέσεις με κάποιες χώρες λόγω θεμάτων δικαιωμάτων του ανθρώπου σε αυτές αλλά και το πως η, ε, το εμπόριο έχει επιπτώσεις στην κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τώρα, σε σχέση με το αντίτιμο, το, στη σωστή τιμή που πρέπει να καταβάλλεται στο εμπόριο. Είναι θέματα που πρέπει να αξιολογούνται σε συμφωνίες και με τα δικαιώματα του ανθρώπου. Και έτσι να δούμε σε σχέση με τις συμφωνίες αυτές τις δυσχέρειες που τίθενται. Και η Επίτροπος Συρία Μάλμστρομ θα υποβάλει προτάσεις από ό,τι γνωρίζω πώς ε, οι ρήτρε ανάπτυξης θα μπορούν να εισαρθούν στα θέματα εμπορίου. Αυτό πάντα είναι ένα ζήτημα. Προσφέρουμε κάτι το δίκαιο ως προσφορά σε αυτές τις χώρες ή κοιτάζουμε μόνο ιδιωτελώς τα δικά μας συμφέροντα. Θα πρέπει να το δούμε αυτό, όρους και προϋποθέσεις και σε σχέση με τα μη δασμολογικά εμπόρια, ε, εμπόδια, διότι αν το προσεγγίσουμε με αυτόν τον τρόπο η προσέγγιση είναι ε, κάνουμε συμφωνίες με αυτές τις χώρες της Αφρικής, ας το λάβουμε υπόψη να μην ε, ξεπερνάμε τα όρια και υπερβάλλουμε. Θα βρισκόμαστε σε λάθος πορεία όμως αν κάναμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για τα, τις ρήτες του των δικαιωμάτων του ανθρώπου, να δώσουμε συνέχεια λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο. Κάποια θέματα Υπάρχουν διαφορετικές ρήτρε για τα δικαιώματα του ανθρώπου σε διαφορετικές περιφερειακές συμφωνίες. Διαρωτώ με, ο κύριος Βάουτερς ή ο κύριος Λότζ θα μπορούσαν να μας δώσουν κάποιες επεξηγήσεις γιατί θεωρείτε εσείς ότι αυτό είναι κάτι θετικό ή όχι και αυτό σε σχέση με μια οικουμενική διακήρυξη όπως για την οικουμενική διακήρυξη για τα δικαιώματα του ανθρώπου και για τις διαφορετικές αυτές ε, πτυχές ε, τι θα κάνουμε στο μέλλον Πώς θα μπορέσουμε στο μέλλον να επιβάλλουμε το σεβασμό αυτών των ρητρών και να μην εκφυλιστεί το θέμα σε μια πολιτική συζήτηση απλώς διότι με τη συμφωνία του Κοτονού όταν ξεκινά ένας πολιτικός διάλογος δεν ξεκινά για τις ρήτρες για τα δικαιώματα του ανθρώπου χειροπιαστά αλλά υπάρχουν ιδιωτέλειες πολιτικές και διεξάγεται ένας τέτοιος διάλογος. Όταν λοιπόν υπάρχει έναρξη κάποιου τέτοιου διαλόγου πρέπει να τα λάβουμε αυτά υπόψη. Αλλά για καθημερινές περιπτώσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου δεν είναι κάτι το ενδιαφέρον και έτσι δεν προσεγγίζονται με πρώτη προτεραιότητα. Και πώς θα μπορούσε ο πρέσβης του Μαυρικίου να τοποθετηθεί. Θα ήθελα να στραφούμε και σε εκείνο το τμήμα των δικαιωμάτων του ανθρώπου που δεν αφορά μείζωνα θέματα όπως την εργασία των παιδιών για παράδειγμα, αλλά για σας, για τη δική σας περιφερειακή συμφωνία για την ανάπτυξη στο εμπόριο, μπορείτε να μας πείτε πώς διασφαλίζετε ότι με τους φόρους θα μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εσείς έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ για τη διεξαγωγή αυτής της ακρόασης. η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι μπόρεσα να ακούσω όλους που παρενέβησαν. Θα ήθελα να κάνω τρεις ερωτήσεις πιο συγκεκριμένες. Η πρώτη. Νομίζω ναι ότι είναι ε, πολύ σημαντικό να εντάξουμε ένα κεφάλαιο για τα δικαιώματα του ανθρώπου μέσα στο κεφάλαιο της αηφορίας ε, για τις εμπορικές συμφωνίες. Πιστεύω ότι το εμπόριο ποτέ δεν είναι αυτός σκοπός και να γίνεται εμπόριο ε, όσον αφορά τις ε, συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Δεν μπορούμε λοιπόν να δεχόμαστε να παράγονται προϊόντα ε, που δεν θα παράγονται με το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε συστήματα αξιολόγησης, παρακολούθησης. Πώς τα κεφάλαια που εντάσσονται υπάρχει πρόοδος για τα δικαιώματα του ανθρώπου και υπό αυτό το πρίσμα και προσέγγιση θα ήθελα να κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Επεσήμανε ο πρέσβης του Μαυρικίου, του Μαυρικίου ότι υπάρχουν και άλλοι πρωταγωνιστές ε, που συμμετέχουν στις εμπορικές πτυχές ε, στα εμπορικά θέματα στην Αφρική. Θα ήθελα να γνωρίζω αν σε αυτές υπάρχουν κάποια κεφάλαια που θα λαμβάνουν υπόψη την αηφόρο ανάπτυξη σεβόμενη σε, πάντα υπό το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου διότι σε σχέση με τις ε, ε, εμπορικές προϋποθέσεις για τις δίκαιες τιμές που πρέπει να ε, ισχύουν πρέπει να δούμε αν όλα αυτά τηρούνται ή όχι. Η άλλη ερώτηση που θα ήθελα να διατυπώσω πώς αξιολογείται την ένταξη των δικαιωμάτων της ισότητας των γυναικών, της ισότητας των φίλων σε όλα αυτά. Είναι σημαντικό και το δικαίωμα στην παιδική ηλικία. Να μην ξεχνάμε όμως και τα θέματα των γυναικών, ιδιαίτερα στις χώρες που πλήττονται ιδιαίτερα από τη φτώχεια και τη βία. Γι' αυτό θα ήθελα να ακούσω την αξιολόγησή σας σε σχέση με αυτή την πτυχή του φίλου και της ισότητας. Ευχαριστώ. ευχαριστούμε. Ο Χέλμουτ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω τους πραγματογνώμενες, πραγματογνώμονες, διότι ο περίπλοκος και σύνθετος χαρακτήρας των θεμάτων, όπως εκφράζεται και όπως είναι δεδομένος, καλύπτεται. Τώρα, για τη συνάδελφο Αργεντίνη, σε σχέση με το θέμα το οποίο τέθηκε, τι είναι για μας τα δικαιώματα του ανθρώπου. Ένα θέμα το οποίο ως κριτήριο απλά και μόνο θα το εγκρίνουμε και τέρμα ή πρέπει να κάνουμε λόγο για την εμπορική μας πολιτική σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ώστε να υπάρξει ανάπτυξη μιας κοινωνίας προς αυτή την κατεύθυνση ώστε οι πολίτες, οι άνθρωποι από την εργασία τους, από την πώληση των προϊόντων τους και την ε, ζωή τους να μπορούν να επιβιώσουν και να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να μπορούν να ευημερήσουν και για την παραγωγή την οποία θα διαμορφώνουν και για τις μελλοντικές γενναίες. Τίθεται το θέμα λοιπόν των δικαιωμάτων του ανθρώπου που δεν είναι καθόλου απλό ως ζήτημα για να ε, το αξιολογήσουμε και να το προωθήσουμε σε σχέση και με τη χάρτα των, δικαιωμάτων του ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών στις σχέσεις μεταξύ των κρατών χάρτα στην οποία με σαφήνεια καθορίζονται ποια δικαιώματα ως δικαιώματα του ανθρώπου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να προάγονται. Και με την χάρτα και την επικύρωση και όταν κάνουμε λόγο για τις ρήτρε για τα δικαιώματα του ανθρώπου σε εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει με κάθε συνέπεια να αναφερόμαστε στις διεθνώς αναγνωρισμένες βάσεις σε αυτή τη σχέση μεταξύ μας στις διεθνείς σχέσεις. Και τώρα το ερώτημα προς τους πραγματογνώμονες υπό το δικό μου πρίσμα, η δική μου προσωπική ερώτηση. Θέλουμε να είναι εφαρμοστέα και δεσμευτικά αυτά τα μέσα σε μηχανισμούς για τις εμπορικές συμφωνίες με ίδια ευθύνη ώστε να μπορούν με υποχρέωση που θα αναλαμβάνουμε εμείς αναγνωρίζοντας το δεσμευτικό τους χαρακτήρα να τα κατοχυρώνουμε. Δηλαδή θα δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό εμείς οι ίδιοι μέσω των εμπορικών συμφωνιών που θα στοχεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλο σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω. Το κριτήριο της συμβατότητας. Αυτό αναφέρθηκε ήδη σε σχέση με συμφωνία Κοτονού και τη συνεκτικότητα. Πολλά συγκεκριμένα στοιχεία σε σχέση με τον ΠΟΕ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και θέματα που δεν κατοχυρώνονται επαρκώς. Εγώ είμαι εισηγητής σε σχέση με την κοινότητα των Ανατολικοαφρικανικών κρατών. Το ερώτημα που τίθεται είναι αυτή η συμφωνία συνάδει, ευθυγραμμίζεται με τις άλλες διεθνείς δομές που ανέφερα πιο πριν ε, διαφορετικά και σε αυτό ανήκει τρίτον και το θέμα της, ε, το ζήτημα που είναι πώς θα αξιολογήσουμε τη δράση μιας ε, επιβεβλημένης υποχρεωτικής πρόσβασης στην αγορά που θα ρυθμίζεται με αυτόν τον τρόπο. Και τι θα κάνουμε, θα στοχεύουμε στην αηφόρο ανάπτυξη με αυτά τα μέτρα για αυτή τη χώρα αυτή θα ήταν η γέφυρα που θα έπρεπε να δημιουργηθεί για την τήρηση και τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αυτή η προσέγγιση εγκάρσια ή οριζόντια πόσο δεσμευτική ισχυρή μπορεί και πρέπει να είναι και υπό αυτή την πτυχή να αξιολογείται. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, αγαπητοί συνάδελφοι, σιγά σιγά αρχίζει να πιέζει ο χρόνος διότι α, όλο και περισσότεροι συνάδελφοι ζητούν να παρέμβουν. Παρακαλώ να είσαστε πολύ σύντομοι, διότι πράγματι και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε να ακούσουμε την τοποθέτησή της και να δώσουμε και την δυνατότητα στους πραγματογνώμονες να απαντήσουν και εκείνοι. Φεράντ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ε, εθνική εορτή στη Γαλλία και βάλα την γραβάτα με τα χρώματα της χώρας μου έχουμε, υπερασπίζουμε τα, γαλλικά δικαιω... τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Γαλλία όπως ξέρετε αλλά εγώ πιστεύω ότι εδώ βρισκόμαστε εκτός του συναγωνισμού επί του θέματος αυτού Σίγουρα έχουμε καλύτερα θέματα να ασχοληθούμε από τις υποθέσεις άλλων κρατών. Δεν καταλαβαίνω πώς λειτουργεί αυτή η ε, κάθετη διπλωματία. Πρέπει να σεβόμαστε την κυριαρχία των κρατών. Δεν έχουμε να δώσουμε κανένα μάθημα σε κανέναν. Ειδικότερα εδώ στην Ευρώπη, σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου ξεκινήσαμε, ανοίξαμε το 17ο κεφάλαιο από τα 32 με την Τουρκία και πιστεύω ότι αντί να κοιτάμε τι γίνεται στην Ιπποσαχαριαφρική, καλύτερα να δούμε τι γίνεται με την Τουρκία. Την Τουρκία που σήμερα καταλαμβάνει ένα κομμάτι ενός ευρωπαϊκού κράτους της Κύπρου η Τουρκία που ανοίγει τα σύνορά της ε, για να παρέχει προμήθειες στην ΤΑΣ και να δημιουργεί προβλήματα στην ευρωπαϊκή διπλωματία. Όλα αυτά με οδηγούν στο να πω κύριε Πρόεδρε ότι πρέπει να κρατήσουμε κάποια απόσταση από αυτά τα θέματα και να αποφεύγουμε τις συστάσεις. Ασχοληθείτε, έχω να πω κυρίως, περισσότερο με τους Ευρωπαίους που βρισκόνται υπό απειλή από την TTIP που αποτελεί πραγματική απειλή για τα έθνη και για την εθνική ταυτότητα του κάθε κράτους. Ευχαριστώ. Äh, η κυρία Φορέντσα. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Τρει ερωτήσεις. Ε, η πρώτη αναφέρθηκε ήδη κατά κάποιον τρόπο από άλλους συναδέλφους πριν από μένα. Αφορά τη δυνατότητα αξιολόγηση του αντικτύπου του ζητήματο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όχι μόνο όσον αφορά τι ρητές αρισιμότητας αλλά και όσον αφορά τι συνολικέ επιπτώσει των ε, συμφωνιών οικονομική εταιρική σχέση. Δηλαδή αν τελικά, μήπω τελικά η συμφωνία ουσιαστικά εφαρμόζει κάποια ε, νέα επικαιοκρατία ε, που επηρεάζει και τα δικαιώματα των ατόμων, τα δικαιώματα στη γη, τα περιβαλλοντικά δικαιώματα. Ουσιαστικά επιδεινώνεται μήπω η κατάσταση λόγω αυτών των συμφωνιών. Ε, ε, Η δεύτερη μου ερώτηση αφορά το θέμα του πώς αξιολογούνται τα αποτελέσματα. Αναφέρθηκε ήδη από την συναδελφή. Το θέμα του φίλου. Πώς επηρεάζει. Λαμβάνεται υπόψη το φίλο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό ήταν το δεύτερο θέμα. Το τρίτο θέμα είναι πιο πολιτικό. Εμείς μιλάμε για εμπορικές συμφωνίες, όπου οι συμβαλόμενοι έχουν ε, οικονομικό βάρος τελείως άνισο, έτσι, διαφορετικό. Υπάρχουν ε, φόρμουλες, δηλαδή διαφορετικές Υπάρχει ας πούμε το δίκαιο του ασύλου, ας πούμε, ε, είναι μία ε, προϋπόθεση που μας δεσμεύει. Θα μπορούσε αυτό να ε, συμβαίνει αυτό στο εμπόριό μας. Νομίζω ότι υποδηλώνει και μία επιθετικότητα, ας πούμε, της Ευρώπης που πλήττει και κάποια δικαιώματα στις χώρες αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να αμφισβητήσω, δεν θέλω να αμφισβητήσω ότι στην σημερινή συζήτηση μια ιδιαίτερα σημαντική παρατήρηση ακούστηκε. Είπε ο πρέσβης του Μαυρικίου ότι το δικαίωμα στην ανάπτυξη είναι και αυτό ένα δικαίωμα του ανθρώπου. Είναι και αυτό δικαίωμα των ανθρώπων και το 2015 το τρέχον έτος είναι έτος ανάπτυξης όπως έχει διακηρυχθεί. Και όλα αυτά τα οποία συνδέονται με τις εμπορικές μας σχέσεις με τις χώρες αυτές, τις αφρικανικές χώρες, όλα αυτά θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής φέτος το 2015, διότι η Αφρική είναι μια ήπειρος που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα ανάπτυξης. Αλλά επίσης έχει και πολλές πολεμικές σειράξεις και συγκρούσεις και υπάρχουν συγκεκριμένα ειδικά προβλήματα για τα δικαιώματα του ανθρώπου στις αφρικανικές χώρες. Αυτά ως εκ προημίου προκατακτική παρατήρηση. Και μία άλλη παρατήρηση ακούστηκε, ένα σχόλιο από πλευρά των προλαλισάντων και αυτό ήταν, αναφέρθηκε ότι η συμφωνία στο πλαίσιο λέει του ΠΟΕ, οι συμφωνίες που συνήφθησαν στο πλαίσιο του ΠΟΕ Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου ήταν καλύτερε και πιο αναβαθμισμένε από ότι οι εμπορικέ συμφωνίε που έχουμε εμεί ενώπιόν μα. Ποια είναι η τοποθέτηση αυτή και γιατί την κάνετε. Γιατί θεωρείτε ότι είναι καλύτερε οι συμφωνίε του Διεθνού Οργανισμού Εμπορίου. Αναφέρεστε μόνο στα προτερήματα και πλεονεκτήματα που απορρέουν για το εμπόριο από αυτό το εμπορικό πλαίσιο ή λαμβάνετε υπόψη και την επιπλέον συγκεκριμένη ρήτρα όπως ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου σε σχέση με τις δικές μας συμφωνίες. Σε τι ακριβώς αναφέρεστε και πώς τα αξιολογείτε, μια και υπήρξε αυτή η κριτικού χαρακτήρα, με κριτικό πνεύμα αξιολόγηση. Εμείς φταίμε. Ποιοι οι εμπλεκόμενες χώρες ε, με τις οποίες συνάπτουμε συμβάσεις. Η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει και το αναφέρει ότι η κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου πρέπει ξεχωριστά να λαμβάνεται υπόψη και να αξιολογείται για τις σχέσεις με τους εταίρους μας με τους οποίους συνάπτουμε τέτοιες συμφωνίες άσχετα αν πρόκειται για πολιτικές συμφωνίες ή εμπορικές συμφωνίες Ευχαριστώ uh, Κυρία Βεργία Ζητώ συγγνώμη Πρόεδρε Θα είμαι τάχιστη Το θέμα που τίθεται είναι ποια είναι η θέση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις ευρωπαϊκές πολιτικές και κυρίως στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν όλο και περισσότερες συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. Καθαρό εμές θα έλεγα. Και η αναπτυξιακή βοήθεια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνεται όλο και περισσότερο. Και είμαστε πολύ μακριά από τους στόχους που είχαμε θέσει πριν από 10 χρόνια. Είχαμε πει 0,7 του ΑΕΠ και έχουμε φτάσει στο 0,29. Πρέπει να είμαστε συνεπεί. Το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα του προβληματισμού μα. Και εγώ έχω τι ίδιε ερωτήσει. Οι συμφωνίε του ΠΟΕ σε τι είναι καλύτερε, α πούμε, από τι συμφωνίε οικονομική εταιρική σχέση, καταρχήν. Δεύτερον, οι Ηνωμένε Πολιτείε σέβονται περισσότερο ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα στις συμφωνίες. Πώς το κάνουν αυτό. Θέλουμε να ακούσουμε συγκεκριμένα πράγματα και εμείς πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Τρίτον, όλοι όσοι δουλεύουν σε αυτά τα θέματα ξέρουν ότι οι ρήτρε για τη δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιωμάτων είναι προσχηματικές. Θα ήταν καιρός, νομίζω, είναι και η ώρα, να κάνουμε πραγματική αξιολόγηση των ρητρών αυτών. Και τι γίνεται με τους άλλους εταίρους. Μιλήσαμε για τη ΣΥΠΑ, αλλά η Ινδία και η Κίνα τι κάνουν. Στις συζητήσεις που έχουμε με αυτές τις χώρες, το θέμα της καλύτερης τιμής δεν είναι αυτό που πριτανεύει τελικά. Επίσης, εγώ θεωρώ ότι τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα είναι πολύ σημαντικά και εκεί στον πυρήνα αυτό βρίσκεται το θέμα των εργασιακών δικαιωμάτων και των συνθήκων εργασίας, τι ρόλο παίζουν οι συνθήκες του ΟΗΤΕ, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Το θέμα της αξιοπρεπούς εργασίας, το θέμα της παιδικής εργασίας, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε για να έχουμε κάποια ελάχιστα, ε, έναν ελάχιστο κοινό παρανομαστή. Και αυτό θα πρέπει να είναι μία ρήτρα ε, η οποία μπλοκάρει. Η, η κυρία Βαλενθιάνου, κάποιε ερωτήσει. Όχι ερωτήσει, θέλω να πω δύο πραγματάκια απλώς. Τίποτα άλλο και μετά κλείνει η συζήτηση. Βρισκόμαστε στην καρδιά του προβλήματος, έτσι. Στην ουσία του ρόλου μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο. Και εδώ υπάρχουν, όπως φαίνεται, τεράστιες ε, αντιφάσεις και τρομερή αναντιστοιχεία. Τι κάνουμε, υποτίθεται. Από τη μία, προσπαθούμε να διατηρήσουμε ρήτρε στη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όμως συχνά μία απλή συμφωνία στις ρήτρε αυτές ε, αμφισβητεί τη δυνατότητα εξαγωγή, δηλαδή μείωση της στόχιας τον 21ο αιώνα θα πρέπει να ξαναδούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρώτα τα ανθρώπινα δικαιώματα και μετά το εμπόριο. Και ξέρω, δεν είναι εύκολο κάτι τέτοιο, αλλά εάν δεν το κάνουμε, μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι επιπτώσεις έχουν οι δράσεις μας στις τρίτες χώρες. Εάν δεν αξιολογούμε αυτά που, γίνονται, τότε τουλάχιστον ας μην είμαστε υποκριτές και α κάνουμε απλώς καθαρόενε εμπορικές συμφωνίε και τίποτα άλλο. Να μην προσποιούμαστε ότι κάνουμε κάτι άλλο. Αυτή η θέση που θέτουμε εδώ, εάν δεν υπάρξουν προσαρμογές, αν δεν αλλάξουμε τις ε, εμπορικές ή πολιτικές σχέσεις με τις τρίτες χώρες, και εδώ δεν πρόκειται να δώσουμε, δεν θέλουμε να δώσουμε δικαιώματα, να είμαστε έτσι, συγκαταβατική κτλ. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι καθολικά, έτσι, και αφορούν όλους. Θέλω να προσθέσω και εγώ, λέει ο δύο πράγματα. Συζητήσαμε λιγάκι την εφαρμογή. Οι εμπειρογνώμονε θα μπορούσαν να μου δώσουν μία συμβουλή. Ποιοι είναι οι φορεί που μας, οι παράγοντες μάλλον που εξασφαλίζουν την εφαρμογή. Επίση, εσεί που κριτικάρετε τι συμφωνίε οικονομική εταιρική σχέση, ποια είναι η καλύτερη εναλλακτική για να βελτιώσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, αν όχι μέσω αυτών των συμφωνιών. Και πριν ξαναδώσω το λόγο στου ε, εμπειρογνώμονε, θα δώσω το λόγο καταρχήν στη Σάντρα Γκαλίνα, στην Κομισιόν, από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Καλημέρα. Σα ευχαριστώ που μα προσκαλέσατε σε αυτή την ε, πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση. Πραγματικά βρισκόμαστε στην καρδιά του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στον κόσμο. Θα ήθελα να ακούσω, να απαντήσω ε, σε διάφορε ερωτήσει, όπω σε εσά, κύριε Παντζέρη. Δεν κάνουμε συμβασμού με τις συμφωνίες οικονομικής και εταιρική σχέση. Έχουμε μια πλήρη πανοπλία, όχι μόνο με αναφορές στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και σε διάφορα εργαλεία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα που ε, εντάσσονται στι συμφωνίε οικονομική εταιρική σχέσης είναι ουσιαστικό, θεμελιώδε στοιχείο σε αυτέ τι συμφωνίε. Δεν έχουμε κάνει κανένα συμβιβασμό επ' αυτού. Υπάρχουν χιλιάδε αναφορέ ε, στα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλε τι συμφωνίε αυτέ. Οποιαδήποτε συμφωνία και να πάρει, θα δείτε πόσε αναφορέ έχουμε. Έχουμε και αποτελεσματικά εργαλεία για να προασπίσουμε, να προάγουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν θέλω να μπω στην ε, συζήτηση αν τα με αυτά τα εργαλεία, αλλά συμφωνώ με εσά κύριε Μάρτιν ότι θα πρέπει να τι αναζωογονήσουμε αυτέ τι συμφωνίε. Έχω πολλές ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, πολλές κοινοβουλευτικές συνελεύσεις. Εάν μπορούμε να κάνουμε μία μικρή διαφορά στην ε, κοινωνία των πολιτών, σε αυτό ήταν σημαντικό. Ο κύριος Κερτεντάλιν ενδιαφέρεται πολύ για το Μασούγο και το Λαμίνι, οι οποίοι έχουν απελευθερωθεί. Θα είδατε το Twitter. Εμείς το καταφέραμε. Και ο Νικόλα Μπελόνο, ε, Μπελόμο έκανε πάρα πολλές προσπάθειες, μπράβο του, Χρειαζόμαστε μια θετική έτσι, στάση απέναντι στους, εμπορικού ε, στους εμπορικούς εταίρους μας. Έχουμε τα εργαλεία, ε, πρέπει να προσπαθήσουμε όμως κιόλα, γιατί δεν είναι τίποτα εύκολο σε αυτές τις χώρες. Και θέλουμε να είμαστε στο πλευρό αυτών που θέλουν αλλαγή στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και όχι μόνο στα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν κολλάμε μόνο αυτό. Επίσης, να πω ότι θα ήταν άδικο να πούμε ότι αυτές οι χώρες έχουν προσυπογράψει ακροτηριασμένες συμφωνίες. Όχι. Έχουν όλες τις αναφορές σε όλα αυτά που θέλετε, ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Και εντάσσονται μετά αυτές οι συμφωνίες και συνδέονται με την Συμφωνία Κοτονού, που είναι η Συμφωνία Αναφοράς και αφορά όχι μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλα τα υπόλοιπα. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να συμβαίνει ας πούμε στις χώρες αυτές, στο μέλλον. Μόνο και μόνο γιατί τα μέρη προσυπογράφουν σε μια συμφωνία που αναφέρει σε αυτά τα βασικά στοιχεία, δηλαδή νομικό πώ σήμερα υπογράφουμε μια συμφωνία με όλα αυτά τα θετικά στοιχεία, τα θεμελιώδη στοιχεία. Είτε υπάρχει το κοτονού είτε όχι, είτε χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία αυτά τα οποία θα τα έχουμε μέσω του διαδόχου εργαλείου του κοτονού ή μέσω μιας, μιας οποιασδήποτε συμφωνίας θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το άρθρο 2.15 και 2.18 της Συνδίκης Λισαβόνας θα ισχύουν πάντα. Γιατί δεν ε, διαπραγματευτήκαμε template, ένα μορφότυπο, γιατί είχαμε αυτό το υπέροχο μορφότυπο ας πούμε, αλλά γιατί. Γιατί δεν θέλαμε να κάνουμε συμβιβασμού στις αξίες. Γιατί κάποια στιγμή οι διαπραγματεύσεις ήταν πολύ έντονες, με πολλές τριβές. Και καλό το κοτονού βέβαια, ε, γι' αυτό ήταν σημείο αναφορά για του εταίρους μα. Αλλά και για μα και για μένα. Να λέω ότι α, είναι θέσπατο το κοτονού, ούτε ακόμα δεν αλλάζω από το κοτονού. Γι' αυτό λοιπόν συνέχεια παραπέμπαμε στο, στο κοτονού. Ε, γιατί εκεί αναφέρεται η, η εργασία, η παιδική εργασία, το περιβάλλον. Είχαμε μια πανοπλία από εργαλεία που ξεπερνούσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μιλούσαν για βιώσιμη ανάπτυξη κανονικά. Στο μέλλον λοιπόν, οτιδήποτε και να συμβεί με το κοτονού, έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τη Λισαβόνα, να αναθεωρήσουμε τη Συμφωνία οικονομική εταιρική σχέση μέσω τη Β' αναθεώρηση. και εσεί θα μου πείτε γιατί διαπραγματευτήκατε, γιατί διαπραγματευτήκατε με το κεφάλι για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, κανένα κενό. Τα έχουμε όλα τα εργαλεία στα χέρια μα. Αλλά α πούμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, τι γίνεται στο μέλλον μπορεί εκεί να έχω ένα κουμπάκι μονομερό στη δική μου ε, διάθεση, έτσι, που δεν είναι κατά ανάγκη καλό για τις χώρες ΑΚΕ. Σήμερα με τη Συμφωνία ε, Κοτονού έχουμε το διάλογο. Έχουμε την εμπλοκή των εταίρων μας στο μέλλον. Εάν δεν υπάρχει το Κοτονού και επομένως δεν υπάρχει αυτή η εμπλοκή, είμαι πεπισμένη ότι καλό θα ήταν ε, οι χώρες ΑΚΕ να διαπραγματευτούν τα κεφάλαια τα οποία λείπουν από τις ΕΠΑ, από τις Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης. Επομένω, σήμερα είναι όλα εντάξει με το κοτονού, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται μετά το 2020. Το 2020. Κοιτάξτε, δεν έχουμε κάνει συμβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν θα πρέπει ποτέ να κάνουμε συμβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το λέω. Από την άλλη, ό,τι και να συμβεί στο μέλλον, έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε έστω και μονομερό κυρώσει. Που εγώ δεν θα ήθελα βέβαια. Θα ήταν πάντα μια τελευταία καταφυγή. Τώρα, στο, στην κυρία Σαρτζεντίνη και στον, στην κυρία Αρένα και στην κυρία Φορέντζα. Θέλω να δώσω μια απάντηση. Έγινε αυτή η παράθεση ε, των Ηνωμένων Πολιτειών σε συμφωνίες που είναι μη ισορροπημένες. Οι Αμερικανοί αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι εμείς προσφέρουμε ασύμετρες συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης. Συμφωνίες δίνουμε, όπου δίνουμε πολύ περισσότερα στις χώρες αυτές από αυτά που μας δίνουν οι εταίροι μας σε εμά, το οποίο είναι πολύ λογικό. Και αυτή είναι ανισορροπία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε μιλάνε για το Sustainably Hold Trade, όπου τι σημαίνει αυτό, ότι εμεί θα είμαστε πιο ισορροπημένοι, δηλαδή θα έχουμε πιο ε, ισόρροπη θέση απέναντι στου εταίρου. Άρα θέλουμε περισσότερε παραχωρήσει από μέρου του. Αλλά εδώ σήμερα μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και θα σα προσκαλέσω σε μια τεχνική συνεδρίαση όπου θα σα δείξω τι διατάξει. Γιατί είναι, πραγματικά άδικο να λέτε ότι οι εταίροι μα δεν κάνουν ε, αρκετέ προσπάθειε. Έχουν προσυπογράψει το πιο αυστηρό, το πιο όμορφο πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μπορεί άνθρωπο να φανταστεί. Thanks a lot. Ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Παντσέρη. Όχι, δεν θέλω να επαναλάβω κάτι απλά. Να πω ότι την επόμενη φορά θα ήθελα να μιλήσετε πρώτα ώστε να μπορούσαμε να απαντήσουμε στο σελέτε. Ναι, ενδεχομένω θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια τεχνική ενημέρωση και να συζητήσουμε τα πράγματα σε βάθο. Ωραία, δίνω τώρα το λόγο στον Ανδρέα Ρώση από το Τμήμα Ανθρωπινών Δικαιωμάτων. Για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση εδώ σήμερα. Δεν θέλω να επαναλάβω τόσο είπε συναδέλφος κύριε Γκαλίνα από την Κομισιόν. Απλά να επισημάνω ότι φυσικά στο πλαίσιο του άρθρου 21 της συνθήκης καθίσταται σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει ότι θα συμπεριλάβει στην εξωτερική δράση τις αρχές της δημοκρατίας, της οικουμενικότητας των δικαιωμάτων, της ενδιαφερότητας των άνθρωπων, όλα αυτά στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης. Αυτά έχουν επικυρωθεί σαφώς, όπως είπε αρχικά ένας από τους εμπρογνώμονες εδώ. Στη στρατηγική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τη δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2012 και στο σχέδιο δράσης αυτή τη στιγμή που εγκρίνουμε αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο και ξέρετε αυτή τη στιγμή Έχουμε ένα νέο σχέδιο δράσης ε, για το διάστημα 2015-2019 που μελετάμε στο Συμβούλιο όπου αναφέρεται αυτή η αρχή και προβλέπονται συγκεκριμένες δράσεις. Αλλά τώρα όσον αφορά το ζήτημα που συζητάμε εδώ σήμερα για τις ρήτερες ανθρώπινων δικαιωμάτων στις διεθνείς συμφωνίες όλες ε, οι συμφωνίες πλαίσια που έχουν ε, συναυθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1995 συμπεριλαμβάνουν τέτοια ρήτρα αποτελεί ουσιώδες στοιχείο των συμφωνιών και αποτελεί το η απόδειξη της βούλησης των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων να συμπεριλάβει τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εξωτερική δράση. Ποια είναι η βασική αξία αυτής της ρήτρας. Είναι ότι και τα δύο μέρη ε, σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρε ΕΣΥΠΗ δηλώνουν μέσω αυτή τη ρήτρα ότι δεσμεύονται από κοινού για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τη δημοκρατία και του κρατού δικαίου. Και αυτό αποτελεί μια νομική βάση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα δύνατο για οποιαδήποτε από τα δύο μέρη να θεωρήσει ότι αυτά τα δικαιώματα είναι απλά εσωτερικό θέμα. Γι' αυτό το λόγο εμεί, ο Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική τη συμπερίληψη των ρητρών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στι μελλοντικέ διαπραγματεύσει με τρίτε χώρε. Τώρα, όσον αφορά την Κοτονού, η τρέχουσα ΣΟΕΣ με τι χώρε ACP θα λήξει το 2020. Ε, με τη λήξη της συμφωνίας θα γίνει ένας απολογισμός της εταιρικής σχέσης και θα διερευνηθεί ε, το τι θα διατηρήσουμε για το μέλλον στο παγκόσμιο πλαίσιο. Όπως ανέφεραν προ... προηγούμενοι η διαδικασία διαβουλεύσεων ξεκινάει τώρα. Η δημοσία διαβούλευση θα ξεκινήσουμε στου επόμενου μήνε και περαιτέρω συζήτηση θα γίνει με του θεσμού και του εταίρου ECP επί του θέματο. Αλλά αυτό που θα ήθελα να τονίσω εδώ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη από τώρα δεσμευτεί να διατηρήσει το πολιτικό διεκτημένο και ειδικότερα τον πολιτικό διάλογο στις διαβουλεύσεις του άρθρου 96 σε οποιοδήποτε πλαίσιο αξιολόγησης, σε οποιοδήποτε ε, μελλοντικό πλαίσιο και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να συμπεριληφθούν ρήτρε πολιτικέ που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτο δικαίου σε όλε τι συμφωνίε που θα συναυθούν. Και αυτό ισχύει και για τι χώρε ACP και για το μέλλον. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Thanks a lot. Ευχαριστούμε πολύ. Δίνω το λόγο ξανά τώρα στου εμπειρογνώμονε. Ο κύριος Βάιτορς, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Πρώτα, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή τη συζήτηση υψηλού επίπεδου και την εξέταση σε βάθος των στοιχείων αυτών σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται και που οι ισορροπίες και αυτές μεταλλάσσονται και η πολιτική και τα νομικά μέσα και αυτά μεταξελίσσονται. Εν συντομία, για κάποια ερωτήματα που στόχευαν σε μένα για τον εφαρμοστικό χαρακτήρα των ρητρών αυτών ε, όσον αφορά τις ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης ε, και σε σχέση με τη Συμφωνία Κοτονού και σε σχέση με τα θέματα του ότι οι συμφωνίες πρέπει να εφαρμόζονται και να ερμηνεύονται ως θέμα αρχής μέσα από αυτά τα συστατικά του στοιχεία και μέσα υπό το πλαίσιο άλλων συμφωνιών ή διεθνών μέσων που τα ίδια εμπλεκόμενα μέρη έχουν ε, συνάψει σε σχέση με τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις τους. Σε σχέση με όλα αυτά δεν ε, νομίζω ότι να υπάρχει οποιαδήποτε αμφισβήτηση για την εφαρμογή τους. Γιατί υπάρχει διαφοροποίηση τώρα των διαφορετικών ρητρών για τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι κάτι το οποίο εξακολουθεί να είναι γρίφος για μένα και δεν έχει απαντηθεί επαρκώς πρέπει να τύχει περαιτέρω εξέτασης και νομίζω συνδέεται με κάποιες από τις ιστορικές συγκυρίες που διείπαν τα πράγματα αυτά κατά το παρελθόν και που οδήγησαν σε <clears throat> αξιοπρόσεκτες καταστάσεις. Για την κοινότητα των κρατών των Άνδεων έχουμε τη συμφωνία του 2012 με την Κολομβία και το Περού με ισχυρέ ρήτρε για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Για τι άλλε δύο χώρε των Άνδεων όμω, Εκουαδόρ και Βολιβία, έχουμε άλλε διατάξει για τα δικαιώματα του ανθρώπου που είναι διαφορετικέ. Όλα αυτά συνδέονται με την υποεξέλιξη ε, αυτών των θεμάτων ιστορικά και με την προσέγγιση γεωγραφικά κάποιων χωρών. Το να θέτουμε το ερώτημα μήπως δεν θα μπορούσαμε τελικά να κινηθούμε προς μια πιο ενιοποιημένη, εναρμονισμένη κατάσταση όπου τα θέματα αυτά τα οποία θα θεωρούμε ότι είναι θεμελιώδους σημασίας θα πρέπει να προαχθούν και νομίζω ότι πρέπει πολύ πιο πέρα να πάμε από μια απλή αναφορά στα οικουμένα, οικουμενικά δικαιώματα του ανθρώπου και τη διακήρυξη των οικουμενικών αυτών δικαιωμάτων του 1948. Από τότε πάρα πολλά μέσα και μέτρα υιοθετήθηκαν και εξελίχθηκαν τα πράγματα, μην το ξεχνάμε αυτό. Και υπάρχει και μια <clears throat> ε, ένα ολόκληρο θέμα ως θησαυρό ε, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου όλα τα κράτη των Ηνωμένων Εθνών εξετάζονται μέσω του EPR, του Μηχανισμού Επανεξέτασης, πράγμα το οποίο δίνει πολλά στοιχεία όσον αφορά τα μέσα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις επιδόσεις ε, που υπάρχουν. Νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες αναφορές έγιναν στον θεσμό μεταξύ εμπορίου και ανάπτυξης. Και πάλι εδώ η συνθήκη της Λισαβόνα ε, πρέπει να πω ότι μας υποχρεώνει να πάμε πιο πέρα από όλα αυτά και να συνδέσουμε τα διαφορετικά στοιχεία των πολιτικών για να δημιουργηθεί μια καλύτερη κατανόηση και να συνειδητοποιήσουμε ότι τα μέσα αυτά πρέπει να ενταθούν ευρύτερα σε μια εμπορική πολιτική και πολιτική ανάπτυξη και να μπορούν να έχουν στενότερη συνέργεια και συντονισμό μεταξύ τους ώστε να βελτιστοποιήσουμε τα αποτελέσματα τα οποία θα ε, ε, έχουμε ως τελική έκβαση. Και κάνοντας λόγο για τους ε, θεσμικούς μηχανισμούς, τέθηκαν κάποια ερωτήματα, δηλαδή τι θα κάνουμε μετά στη συνέχεια με αυτές τις ρήτρες των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Είναι σημαντικό να δούμε την παρακολούθηση και συνέχεια που δίνεται ή την απουσία εποπτείας και συνέχειας. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν υπάρχει ούτε μία από αυτές τις συμφωνίες που σε σχέση με τους μηχανισμούς ε, να ε, έχει αυτή την πτυχή. Βλέπουμε έναν πολιτικό διάλογο που συνεχίζεται απλά, πολύ σημαντικό μεν αυτό, αλλά όπως ένας από τους ευρωβουλευτές πολύ σωστά ανέφερε, αυτό τι δίνει, δίνει μία ας το πω έτσι επικέντρωση σε καταστάσεις κρίσης, σε παραβιάσεις ή παραβάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου και εξελίσσεται έτσι ένας πολιτικός ε, διάλογος. Το θέμα όμως είναι να δούμε την παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών καθημερινά σε πολλές χώρες, πράγμα που απαιτεί έναν αυθεντικό μηχανισμό εποπτείας και παρακολούθησης και έναν τρόπο να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα θέματα που κινούμε την κοινωνία των πολιτών και όλους τους ενδιαφερόμενους εμ εμπλεκόμενους γύρω από τη στρογγυλή τράπεζα και η συμβατότητα όλων αυτών είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει επί μεγάλο χρονικό διάστημα παραδοσιακά. Έχει εξεταστεί, έχει συζητηθεί και αναλυθεί και μπορεί να δώσουμε συνέχεια στην εξέταση αυτών αλλά πάντα θα είναι η συζήτηση με τους Αμερικανούς που θα διεξάγεται για τα τι απαιτείται για τις ε, εμπορικές συμφωνίες και μέσα στο πλαίσιο των συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Και είναι θέμα το οποίο επαφήνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναλάβει τις, σωστά, τα, ε, τις σωστές δράσεις και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου που βρίσκεται υπό εξέλιξη βλέπουμε ότι ο αναπτυξιακός γύρος, η πρωτοβουλία αναπτυξιακή της ΔΟΧΑ έχει ε, αποτελματωθεί και βλέπουμε ότι εδώ για όλες αυτές τις ε, περιφερειακές συμφωνίες στον 21ο αιώνα πρέπει να ε, αναλάβει τις ευθύνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για να δώσει το σωστότερο πλαίσιο για αυτές. Ευχαριστώ κύριος Λότζ. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Επιτρέψτε μου να κάνω 3,5 ε, σύντομα σχόλια. Το ε, ε, θέμα των ΙΠΑ. Καμιά φορά αξίζει να δούμε τι κάνουν οι ΙΠΑ και πώς προσεγγίζουν οι ΙΠΑ κάποιες από αυτές τις εμπορικές συμφωνίες. Αν δει τώρα τις διατάξεις που υπάρχουν και που επειδή οι ΙΠΑ σε αυτό το πλαίσιο όταν δραστηριοποιούνται έχουν κάποια ε, επιχαίρουν, καμιά φορά όταν βλέπουν ότι ε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τα ίδια ζητήματα και θέλει να βρει κάποια διέξοδο πώς δηλαδή μπορεί να ακολουθήσει την πορεία των ΗΠΑ ε, σε σχέση με αυτές τις ε, περιφερειακές συμφωνίες και συμφωνίες για την ανάπτυξη και το εμπόριο υπάρχει μία διάταξη που είναι οικουμενικά πανομοιότυπη ή συγγενής. Οποιαδήποτε υπαναχώρηση, οποιαδήποτε ε, ανταπόκριση γίνεται πρέπει αυτόματα να ισχύει και για τη ΣΥΠΑ. Δεν υπάρχει καμία ε, ας το πω έτσι ε, ξεχωριστή αντιμετώπιση για το επίπεδο ανάπτυξης ή εξέλιξης οποιασδήποτε χώρας. Πρέπει να εφαρμόζεται αυτή η αρχή και σε σχέση με την τρέχουσα μορφή θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα εφαρμόζονται αυτά σε χώρες που 1% του παγκοσμίου εμπορίου θα μπορούν να, να συναποτελούν. Τρεις παρατηρήσεις για την εφαρμογή για την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών. Ένα θέμα το οποίο τέθηκε από παρέμβαση πιο πριν. Πρέπει να είμαστε σε θέση να έχουμε το θέμα της ε, αηφορίας στην ανάπτυξη επειδή υπάρχουν δεσμεύσεις για επενδύσεις ε, και υπηρεσίες. Και ένα από τα σημαντικά θέματα που πρέπει να αναγνωρίσουμε είναι ότι δεν είναι υπό τους όρους των αναφορών στα δικαιώματα ανθρώπου αλλά και για την αηφορία στην ανάπτυξη δεν έγκυται απλώς στο προήμιο αλλά έχει ε, ξεχωριστό χαρακτήρα στα επιμέρους, στα επιμέρους εδάφια και να λάβουμε υπόψη εδώ και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ε, ε, διατάξεις που πρέπει να είναι σεβαστές. Και αυτό είναι ένα στοιχείο διαφοροποίησης όσον αφορά τις άλλες εταιρικές συμφωνίες εμπορικής, ε, εμπορικών σχέσεων και ανάπτυξης. Και ενώ είναι επαναστατικό ή ε, καινοφανές και καινοτόμο σαν στοιχείο στα χαρτιά, δεν έχει επωφεληθεί από το επίπεδο επαρκούς εφαρμογής όπως ε, θα έπρεπε να είχε επωφεληθεί. Και εδώ αμφότερες οι πλευρές ε, είναι ένοχες και σε σχέση με την ασύμετρη ή μη συμμετρική διαμόρφωση των πραγμάτων το ότι η μία πλευρά επομίζεται περισσότερες ευθύνες, ας το διατυπώσω έτσι, από ό,τι άλλοι, εδώ ελπίζω, ευελπιστώ ότι η Επίτροπος Μάλμστρομ όταν θα συνέθει με τους εταίρους της αύριο θα μπορέσει να τους πει προσέξτε έχουμε μεγάλο, μεγάλη μοχλική, μοχλευτική ικανότητα στις διεθνείς οργανώσεις και στους διεθνείς οργανισμούς θα δώσουμε, ε, θα προτρέψουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα στο, στην διαμόρφωση αυτών των μηχανισμών να σας συνεπικουρήσουν στην φορολογική μεταρρύθμιση ώστε οι διατάξεις που έχουμε όσον αφορά την ε, απάλληψη δασμών ε, και υποχρεώσεων να μην οδηγήσει στην μείωση των φορολογικών εσόδων των χωρών της Καραϊβικής. Τέτοιου είδους προτροπές ε, και κίνητρα χρειάζονται. Και είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτό. Αυτό που έχουμε ως μέσα EDF ε, είναι πολύ θετικά και πολύ επικοδομητικά. Όμως ε, δεν, είναι, δεν έχουν τον ευαίσθητο χαρακτήρα σε σχέση με την χρονική συγκυρία που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και ταυτόχρονα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν ξεχωριστοί παράγοντες που διαμο... Ε, ξεχωριστά αντιμετωπίζουν την περιοχή αυτή της Καραϊβικής και των χωρών της Καραϊβικής. Τρεις, ε, ε, τρία στοιχεία ε, λαμβάνοντας υπόψη το ότι έχουμε μια ελάχιστα ανεπτυγμένη χώρη, χώρα, την IT και να δούμε εδώ την ε, ε, ξεχωριστή αντιμετώπιση της. Δεύτερον, σε σχέση με το υπουργικό πλαίσιο και το ε, συμβουλευτικό πλαίσιο για την παρακολούθηση των διαπραγματεύσεων, αλλά το τρίτο πλαίσιο είναι το FTA, Free Trade of the Americas, ελεύθερο εμπόριο στην Ήπειρο της Αμερικής. Είναι ένα σημαντικό πρότυπο το οποίο Δηλαδή τις εργασίες ε, για μας. Δηλαδή πώς θα πρέπει να διαμορφωθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Ε, έχοντας εξοικειωθεί με αυτό το πλαίσιο έχουμε επίσης και ένα άλλο συμβουλευτικό σώμα το οποίο θα μπορούσε να εμπλακεί σε σχέση με τους μη κρατικούς εταίρους και τρίτον ανανέωση η αναζωογόνηση της τάσης να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τα μεγαλύτερα βιομηχανο, βιομηχανοποιημένα βιομηχανικά κράτη, Καναδά, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με το ποια είναι τα ξεχωριστά του συμφέροντα και πώς θα μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε. Τελική μου παρατήρηση σε σχέση με αυτό το συνολικό πλαίσιο. Αυτή η συζήτηση τι καταδεικνύει, ότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για τη μεγάλη σπουδαιότητα των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε σχέση με αυτές τις εμπορικές ε, συμφωνίες. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Το σημαντικό ζήτημα είναι πώς θα κινηθούμε από την ε, ε, διατύπωση ή ε, το φραστικό επίπεδο σε ένα ουσιαστικότερο επίπεδο δεσμεύσεων, εποπτείας και εφαρμογής και εδώ θα είχα τα εξή επιχειρήματα, ότι έχουμε τρεις επιλογές. Η πρώτη είναι η προσέγγιση των ΙΠΑ. Δηλαδή, να καταλήξουμε στην ε, ολοκλήρωση τη της σύναψης τέτοιων συμφωνιών υπό τον όρο και προϋπόθεση ότι προηγούμενα θα έχουν εγκριθεί και επικυρωθεί διεθνείς συμβάσεις παράδειγμα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Να δούμε δεύτερον σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση προσεγγίζει αυτά τα θέματα και με ποιους όρους και προϋποθέσεις εργασιακά θέματα θα μπορούν να εντάσσονται και να εφαρμοστούν στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών. Και το τρίτο, το πλαίσιο της αναγνώρισης ε, ότι οι σχέσεις ΕΕΑΚΕ είναι τόσο ε, ξεχωριστές ε, επειδή στο συμβατικό πλαίσιο και συμβατικό πλαίσιο όχι μόνο έχοντας μια ε, συμβατική διάσταση για το εμπόριο αλλά και πέρα από αυτήν ένα ολόκληρο, μια πανοπλία μέτρων α, ως εργαλειοθήκη για την παρακολούθηση και συνέχεια σε αυτά. Ευχαριστώ. Έχετε τον λόγο πρέσβη του Μαυρικίου παρακαλώ. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση, ακούστηκαν πολλές ερωτήσεις, δεν νομίζω ότι μπορούμε να τις απαντήσουμε όλες, αλλά σημείωσα τρεις-τέσσερις που θα απαντήσω γρήγορα. Για το θέμα της πραγματικής πολιτικής στην Αφρική. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες στην Αφρική, αυτό είναι αλήθεια. Και μερικοί από αυτούς τους άλλους παίχτες δεν βάζουν προϋποθέσεις καθόλου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Κάποιο ρώτησε αν μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα και αν συμπεριλαμβάνουν θέματα που συνδέονται με την βιώσιμη ανάπτυξη αυτοί οι άλλοι παίκτε, αυτοί οι άλλοι εταίροι. Όχι. Λυπόμαστε και εμεί, όχι μόνο η Ευρώπη δηλαδή, αλλά και εμείς, ε, οι Αφρικανοί. Καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι προς το καλό και προς το συμφέρον της Αφρικής. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Από ευρωπαϊκή σκοπιάς νομίζω ότι υπάρχει μια δυνατότητα να κάνετε κάτι γι' αυτό. Και όπως είπε και ένας ευρωβουλευτής, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Να το αντιμετωπίσετε εσείς οι Ευρωπαίοι δηλαδή. Πώς. Υπάρχουν τα έξυπνα κίνητρα, όπως λέμε, τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν, ούτω ώστε να υπάρχει ε, να δίδεται βοήθεια χωρί όρους, αλλά μια και υπάρχουν αυτές οι ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να έχουμε και μια έξυπνη προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είπε και κάποιος ευρωβουλευτής. Επίσης υπάρχει ανάγκη να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια συνεπής πολιτική. Πολύ συχνά αυτό που βλέπουμε είναι ότι, και αυτό όλοι το συνειδητοποιούμε, ότι υπάρχουν διπλά μέτρα και σταθμά. Ανάλογα με, το, με ποια χώρα έχουμε να κάνουμε, αν είναι μεγάλη και δυνατή, έχουμε την τάση να κλείνουμε τα μάτια σε σχέση με το τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Ενώ αν είναι μια αδύναμη χώρα, την τζακίζουμε. Αυτά τα δύο μέτρα και σταθμά, αυτές οι ασυνέπειες θα πρέπει να αποφευθούν. Επίση, ανέφερα ότι υπάρχει ανάγκη να δείξουμε ευαισθησία στην τοπική πραγματικότητα. Κάποιο με ρώτησε πόσο χρόνο πρέπει να δώσουμε σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Εγώ να σας ανταπαντήσω. Στην Ευρώπη πόσα χρόνια κάνατε για να κάνετε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Μπορούμε να περιμένουμε ότι κάτι που πήρε δεκά, δεκάδες χρόνια ή και αιώνε για να συμβεί στην, ε, στην Ευρώπη πρέπει να γίνει μέσα σε λίγα χρόνια, σε δύο χρόνια, πέντε χρόνια, δέκα χρόνια στην Αφρική, είναι δυνατόν. Πρέπει να δώσετε χρόνο σε αυτά τα πράγματα. Μια άλλη ερώτηση. Ε, το εμπόριο είπαμε ότι είναι εργαλείο για την ανάπτυξη. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή να απολαμβάνει ο κόσμος τα ανθρώπινα δικαιώματά του αν δεν υπάρχει ανάπτυξη. Και αν συμφωνήσουμε με αυτό, τότε το εμπόριο μπορεί να είναι εργαλείο για την ανάπτυξη. Αν συμφωνήσουμε σε αυτό, θα πρέπει να προσαρμοστούμε ούτως ώστε η ανάπτυξη να συνεχίζει και να ενισχύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και κάτι άλλο, γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα που αφορά άμεσα τον Μαυρίκιο. Εάν δηλαδή οι πολυεθνικές εταιρείε πληρώνουν τους φόρους τους. Η απάντηση είναι καταφατική. Ναι, τους πληρώνουν. Έχουμε εταιρικούς φόρους ε, με συντελεστή 15% στο Μαυρίκιο. Και επειδή υπάρχουν και κάποιε ε, πολυεθνικές ή παγκόσμιε εταιρείε που πληρώνουν και φόρου στη χώρα τη εταιρική έδρα του, σε αυτές τις περιπτώσεις, για αυτές τις χώρες, τους δίνουμε μία πίστοση φόρου έκπτωση φόρου δηλαδή, ούτω ώστε να μας δώσουν ένα χαρτί ε, που θα αποδεικνύει ότι πλήρωσαν χι φόρου, α πούμε, σε αυτέ τι χώρε και άρα κάνουμε μία αφαίρεση. Ε, δίνουμε δηλαδή ε, φορολογική πίστοση ή έκπτωση φόρου 80% υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πληρώσει αλλού τους φόρους τους. Και αυτό το κάνουμε γιατί ε, εμείς υποβάλλουμε τους φόρους μας σε άλλη χρονική στιγμή. Ας πούμε, εμείς υποβάλλουμε το, τις φορολογικές μας δηλώσεις ε, τον Απρίλιο. Ενώ σε άλλες ε, χώρες μπορεί να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις το Δεκέμβριο. Γι' αυτό το δίνουμε λοιπόν αυτό το χαρτί, αυτή τη, φορολογική πίστοση ας πούμε για να δείξουμε ότι έχουν πληρώσει τους φόρους τους εδώ. Ε, και παρόλα αυτά οι φόροι που πληρώνουν εξακολουθούν να είναι υψηλότεροι και το σύστημα είναι ε, πολύ καλύτερο από αυτά που συμβαίνουν σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από αυτά που είδαμε πρόσφατα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο τελευταίο ομιλητή είναι ο κ. Μπερτολό. Αν επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, όπως πρότεινε η κυρία Μαρία Αρένα, θα ήθελα η απάντηση να προέλθει από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού, Μαντούσοκο. αν το επιτρέπετε. Του δίνω τον λόγο, αν το επιτρέπετε, στον κύριο Μαντούσοκο. Αν αποσύρετε την παρέμβασή σας, θα πάρει λοιπόν αυτό τον λόγο για τρία λεπτά. Merci. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μας δώσατε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε αυτή την πολύ διαφορετική συζήτηση. Θα ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Πρέσβης. Όλοι συμφωνούν ότι το εμπόριο δημιουργεί ανάπτυξη και θέσεις εργασίας και ότι υπάρχουν προϋποθέσεις ώστε αυτό να είναι δυνατό. Βρισκόμαστε στην ακριβή χρονική στιγμή όπου δημιουργούμε μια περιφερειακή ζώνη ώστε να επιτύχουμε όλα αυτά. Θεωρώ λοιπόν ότι η χρονική στιγμή και οι προθεσμίες είναι πολύ σημαντικές. Αν πάτε να συγκρίνετε την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στο πλαίσιο των ΣΟΕΣ ε, με τον ΠΟΕ και θεωρείτε ότι ο ΠΟΕ είναι καλύτερος είναι διότι ο ΠΟΕ ε, επιτρέπει εξαίρεση για τις χώρες ε, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει υπάρχουν άλλοι φόροι φόροι 5% για τα βασικά προϊόντα ε, που στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες είναι, φορολογούνται με 0% βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα ουσιώδες ζήτημα για να μπορέσει το πλαίσιο λοιπόν επειδή εγώ θεωρώ ότι οι ΣΟΕΣ είναι ένα πλαίσιο για να είναι ωφέλιμο λοιπόν αυτό το πλαίσιο Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πολλές από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ε, τώρα ολοκληρώνουν τις διαρθρωτικές αλλαγές. Ε, μιλάμε για εμπόριο, λες και η χώρα ήταν αυτόνομη. Ενώ πολλές χώρες ακόμα εξαρτώνται από κάποιες διαπραγματεύσεις με την Παγκοσμία Τράπεζα, με το IMF, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Υπάρχουν ε, σχέσεις ε, στο πλαίσιο της δημιουργικής συνεργασίας που δεν έχουν ληφθεί απόλυτα υπόψη. Αυτό που θεωρούμε λοιπόν εμείς είναι ότι σήμερα, όπως είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΣΟΕΣ είναι για να ευνοήσουν την ε, περιφερειακή ολοκλήρωση. Αυτή η περιφερειακή ολοκλήρωση σκοπό έχει να προστατευτούν τα, τα όπλα ξέρετε είναι για να προστατεύσουμε τα σύνορα αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ένα χρηματιστήριο μια ελεύθερη αγορά διαφανή και οργανωμένη. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το πλαίσιο το οποίο μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ολοκληρώσω λέγοντας επίσης ότι κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται να χρηματοδοτήσει μια μελέτη η οποία στο τέλος λέει ότι δεν υπάρχουν πολλά πλέον η μελέτη αυτή απορρίπτεται Λυπάμαι λοιπόν, που το λέω, αλλά έχουμε και αποδεικτικά στοιχεία που μπορούμε να εμφανίσουμε εδώ. Μιλάμε για μελέτες που έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίες έδειξαν ότι μέσω των όσων μας προτείνεται τα κέρδη είναι λιγότερα από ό,τι αν είχαμε κάνει διαφορετικά. Τώρα όσον αφορά τα δικαιώματα πιστεύω ότι το βασικό δικαίωμα είναι επί μακρόν ο πληθυσμό και το, το κράτο να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Αυτό είναι το πιο βιώσιμο. Πιο βιώσιμο από τι ελευθερίε και τα δικαιώματα που προτείνουμε, όπω κάνετε αυτή τη στιγμή. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Um, Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, από πλευρά μου, κυρίε και κύριοι, να ευχαριστήσω του εμπειρογνώμονε και του συναδέλφου για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση και πιστεύω ότι το ζήτημα της σωστής εφαρμογής της ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της παρακολούθησης της ε, διαδικασίας υλοποίησης θα αποτελέσει στοιχείο κλειδί στις συζητήσεις μας στο πλαίσιο της ΕΠΑ. Τώρα δίνω τον λόγο στην Έλενα για να ολοκληρώσουμε. Όλοι είναι κουρασμένοι και πεινάει πολύ. Ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.